Um, I would like to start. Um, uh, σας ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι είναι πολύ μικρή αίθουσα για να σας χωρέσει όλους. Όμως, ούτως έχουν τα πράγματα. Ίσως μπορείτε να αλλάζετε θέσεις από καιρού καιρών. Εκείνοι που είναι όρθιοι να κάθονται μετά και οι άλλοι να τους παραχωρούν τη θέση τους και να αλλάξει πάλι. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρωτού ε, προχωρήσουμε, αν συμφωνείτε, θα ήθελα να κάνουμε ένα πράγμα το οποίο αφορά τι εργασίε τη Επιτροπή μα. Έπρεπε σήμερα το πρωί να το έχουμε διευθετήσει, δεν το κάναμε, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε κάποιου συναδέλφου, ήθελα να σα ενημερώσω, για το δεύτερο ήμιση τη κοινοβουλευτική μα θητεία. Είχαμε κάποιε αντικαταστάσει και αυξήσαμε και τον αριθμό των ατόμων στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Με τον Γιένς Νίλσον να ξεκινήσω που αύξησε τον αριθμό των συναδέλφων που ανήκουν κιόλας στην σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Γιάννης Νίλσον, ένας παλαιός φίλος όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Βρισκόταν επί χρόνια στην Επιτροπή Περιφερειών. Δεν είναι καθόλου καινούριο λοιπόν. Έχουμε κάποιον που έχει τεράστια πραγματογνωμοσύνη και αυτό είναι πολύ καλά μαντάτα. Καλή είδηση. Στην Άλντε επίση ω ομάδα έχουμε την Βιντσέντσα Γιωβίνε. Παρακαλώ. Τον Βιντσένσο Βιντσέντσο Γιώβινε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και στην ομάδα των Πρασίνων την Άννα Μιράντα. Χαρά να είσαστε πάλι εδώ ανάμεσά μα, να σα έχουμε εδώ. Και θα έλεγα ότι από πλευρά ε, τη γιατί έχουμε τον Φιλίπ Ντεβίγε, δεν ξέρω, παρίσταται ο κύριο. Εν πάση περιπτώσει και ένας ακόμα συνάδελφος πρέπει να πω που αντικατέστησε έναν άλλον και που επανήλθε Γιούνουσο Ομαζή που βρίσκεστε εδώ χαρά για μας να είσαστε ανάμεσά μας ναι α ο Επίτροπος μου είπε ότι και η Εύα Στάντλερ είναι εδώ ανάμεσά μας καλό που σας βλέπουμε και είσαστε εδώ καλώς ήρθατε Λυπούμε, είναι και κάποιο άλλο που δεν ανέφερα, κάποιο καινούριο, αν υπάρχει να μου το πείτε ποιο είναι. Όχι, ο Ούγγρος συνάδελφος Τσάμα Σέβεντι δεν είναι εδώ παρόν. Εντάξει, και αναπληρωτής η Βαρυπάδο νομίζω που αναπληρώνει ως καινούριο μέλος ε, συνάδελφο. Και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τις επίσημες εργασίες μας. Έχουμε τον Επίτροπο ανάμεσά μας. Πολύ καλό που σας ξαναβλέπουμε για πρώτη φορά εφέτος. Ε, σας εύχομαι καλή χρονιά. Επίσημα σας ξαναβλέπουμε για πρώτη φορά. Ναι, συναντούμε πολλούς. Ε, ευχαριστούμε για το ανοιχτό πνεύμα και την προθυμία σας να μας συναντήσετε και να συζητήσετε μαζί μας. Σήμερα θα θέλαμε να σας ακούσουμε προσεκτικά να τίνουμε δίκο νους γιατί θα θέλατε να σχολιάσετε για τις διαπραγματεύσεις για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Και ως ήθιστε θα ξεκινήσουμε με την εισαγωγή του Επιτρόπου και μετά και πάλι ως ήθιστε θα ακολουθήσουν σχόλια, ερωτήσεις, παρεμβάσεις που θα προέρχονται από τους συντονιστές και τα μέλη τους υπολείπου, τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ Ντανούτε. Θα ήθελα να δραχθώ λοιπόν της ευκαιρία, ιδιαίτερα σε σένα Ντανούτα, αλλά και στους άλλους συναδέλφου που επανεξελέγησαν, ήθιστε, είναι παράδοση στο σώμα, κατά το ίμιση της περίοδου, της κοινοβουλευτική περίοδου, να υπάρχει επανεκλογή, να γίνονται νέε εκλογέ, ώστε να διασφαλίσετε η συνέχεια των εργασιών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και αυτό είναι πολύ θετικό, θα λέγα εγώ ιδιαίτερα στην περιφερειακή πολιτική, οποιαδήποτε μορφή συνέχειας είναι κάτι το ξεχωριστά θετικό και σημαντικό, ιδιαίτερα για την υλοποίηση, την εφαρμογή των πολιτικών μας και των σχεδίων μας και γιατί πραγματικά πρέπει να καταλήξουμε στην αφετηρία από την οποία θα ξεκινήσουμε, διότι είναι χαρμόσυνο τις τελευταίες ε, μέρες και εβδομάδες η διαρθρωτική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όλων, διότι τώρα για την διαθεωτική πολιτική. Πολλοί πιστεύουν ότι το σύνολο των οικονομικών προβλημάτων της Ευρώπης μπορεί να επιληθεί με αυτή την πολιτική. Μπορούμε να συνεισφέρουμε με τη διαθεωτική πολιτική βέβαια και να συνεισφέρουμε στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε όμως τα πάντα. Και πέρα από αυτό, εξ ονόματος όλων νομίζω μπορώ να πω ότι η διαθεωτική πολιτική αφεαυτής είναι μια πολιτική για την ανάπτυξη εξαρτάται με ποιο, πόσο ευφυή τρόπο θα χρησιμοποιούνται τα μέσα. Η στόχη όμως, η στοχοθέτηση είναι σαφής ότι μέσω των κονδυλίων των διαθροτικών ταμείων θα προάγεται η ανάπτυξη, θα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης ή θα διασφαλίζονται θέσεις απασχόλησης. Για να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση για την χρήση των κονδυλίων πέρυσι, 2011, διότι είχαμε ρεκόρ, έτος ρεκόρ απόλυτα. Συνολικά 32 δις ευρώ κατα, ε, πληρώθηκαν καταβλήθηκαν από πλευρά ε, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξη 24,8 ε, από το Ταμείο Συνοχή 6, συν 6,5 σε σχέση με το 2010. Κατά 6,5 δις αξήθηκαν τα κονδύλια αυτά σε σχέση με το 2010. Αυτό ανταποκρίνεται στην εξέλιξη αυτών των πολιτικών και με βάση τις δικές σας αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης και πριν από την αλλαγή του έτους είχαμε 350 πρόσθετ στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και εντωμεταξύ έχουμε και 600 εκατομμύρια ευρώ καταβολή στην ε, Πορτογαλία. Η υλοποίηση των πολιτικών μας λοιπόν αυτών βαίνει με καλούς ρυθμούς και ανταποκρίνεται στις αποφάσεις και ανάγκες. Το 2012 θα πρέπει να είναι έτος εκτέλεσης και εφαρμογής ε, των ηλυμένων αποφάσεων. Θα πρέπει να καταδείξουμε, να αποδείξουμε ότι τα κονδύλια επαρκώς ε, θα αντληθούν και θα χρησιμοποιηθούν θετικά. Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε πολιετή πείρα. Πότε ακριβώς οι πληρωμές, οι απαιτήσει πληρωμών υποβάλλονται και εξοφλούνται. Δεν είναι ασυνήθιστο κατά τα τέλη του έτους να έχουμε υψηλότερο ποσοστό αυτών των υποθέσεων. Τον Δεκέμβριο όμως 18% ε, του συνολικού προϋπολογισμού ε, κατεβλήθη, πληρώθηκε. Και αυτό επειδή ο σχεδιασμός, η σχεδιασιμότητα εντός εισαγωγικών, να την αποκαλέσω έτσι, παρόλες τις ιστορικές, την, την ιστορική μας πείρα ή εμπειρία ε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Η πρόληψη λοιπόν πρόνοια πρέπει να ληφθεί για την ρευστότητα που πρέπει να διασφαλίζεται. Το λέω αυτό επειδή τι λένε και κυκλοφορούν κάποιε φήμε ότι τα μη χρησιμοποιημένα ταμεία των διαθετικών ταμείων θα χρησιμοποιηθούν τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια για άλλη στοχοθέτηση, για άλλου σκοπού. Έτσι λοιπόν τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια όταν δεν έχουν δεσμευτεί, ίσως μπορεί να, να το κάνουν αυτό. Το 2010 προς 2011 είχαμε 30 εκατομμύρια κατά μέγιστο ποσό που δεν είχε δεσμευτεί. Αν 25% από αυτά τώρα ε, θα ήθελαν ευρωπαϊκά να ε, επαναχρησιμοποιηθούν, πάλι δεν θα υπαρκούσαν πλήρως. Το λέω αυτό διότι είναι σημαντικό τουλάχιστον από τον κύκλο των ε, διαφορετικών πολιτικών ε, να υποβληθούν ε, προτάσεις πώς θα έπρεπε να προχωρήσουμε παραπέρα. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό η ποιότητα των σχεδίων να μην βρίσκεται, να μην χωλαίνει να μην ε, ε, έχει διαφορές από το επίπεδο που πρέπει να διασφαλίζεται. Και εκεί που πρέπει να ε, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις και τροπολογίες στα σχέδια και προγράμματα, εκείνα που λειτουργούν καλά θα πρέπει να συνεχιστούν. Εκείνα που δεν λειτουργούν καλά και δεν έχουν τέτοια στρατηγική σημασία θα μπορέσουν με ελαστικό ευέλικτο τρόπο να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει αυτά για τις εξελίξεις αυτές. Και κατά την έναρξη του έτους η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα ενημερώνεται για τις τρέχουσες εργασίες και πώς έχουν εξελιχθεί και διαμορφωθεί τα πράγματα. Και με το σκηνικό μια και εσεί ω κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι εγκρίνετε τα δημοσιονομικά κονδύλια στο πλαίσιο του προπολογισμού ετήσια και για τι προτάσει που υποβάλλετε για τον προπολογισμό. δεν είναι αυτό τίποτα άλλο παρά η ομαδοποίηση και η επιμέρου ε, έγκριση κονδυλίων ανάλογα με τι ανάγκε ρευστότητα που υπάρχουν τις αναγκαιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και όταν έχουμε περικοπές κονδυλίων αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά το ότι τα, ότι τα συμφωνηθέντα κονδύλια δεν θα πληρώνονται στις χώρες που τα έχουν ανάγκη, παρότι έγκαιρα έχουν, θα έχουν αποσταλεί ή αποστέλλονται αιτήσει και αιτήματα. Και στο τέλος, τέλος όταν έχουμε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις πρέπει στο τέλος να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε με τα κονδύλια που έχουμε διαθέσιμα στις ανάγκες μας ε, πολιτική συνοχή μέχρι το 2020 ω στρατηγική. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλου του συμμετέχοντε για το έργο και την, από την παρουσίαση των προτάσεών μα ε, αρχέ Οκτωβρίου του προηγουμένου έτου να σα ευχαριστήσω. Τι έγινε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας αναφέρω ότι όπως αναμέναμε, η Πολωνική Προεδρία έστρεψε με ιδιαίτερη προσοχή το βλέμμα της σε αυτό το πεδίο πολιτικής. Κατέβαλε έντονες προσπάθειες και η συζήτηση στο Συμβούλιο προήχθη, πρόοδευσε και μάλιστα είχαμε και ένα πρώτο κείμενο συμβιβαστικό το οποίο υπευλήθη προς έγκριση το Δεκέμβριο. Και από πλευρά του Συμβουλίου διεξήχθησαν συζητήσεις μήπως ήταν λέει πιο πρώιμη, πολύ πρώιμη αυτή η χρονική στιγμή. Όμως καταδείχθηκε ότι κάποια κράτη μέλη και ιδιαίτερα η Πολωνική Προεδρία σε αυτές τις διεργασίες αυτό το έγγραφο, αυτή την πρόταση με το θέμα της ε, στρατηγικής, ε, του στρατηγικού προγραμματισμού και της θεματολογικής επικέντρωσης και στοχοθέτησης ασχολήθηκε. Είμαι ευγνώμων για το ότι η Δανέζικη Προεδρία με την ίδια προσοχή στρέφεται στην προσπάθεια συνέχισης αυτών των, συνέχειας αυτών των συζητήσεων και υποβάλλει ένα φιλόδοξο σχέδιο και στο πλαίσιο της Δανέζικης Προεδρίας ιδιαίτερα γίνεται λόγος για στοχοθέτηση στη διαχείριση, management και ελέγχους. Ε, και από πλευράς του Συμβουλίου για τον δικό μας τομέα πολιτικών ήδη πάνω από 100 ώρες ε, έγιναν διαπραγματεύσεις για τις διαθρωτικές δράσεις, structural action και είχαμε ένα άτυπο, ας το πω έτσι, επίπεδο ομάδας εργασίας, υπουργικής ομάδας εργασίας ε, με διαβουλεύσεις για αυτά τα θέματα και θα συνεχιστεί αυτή η διαβούλευση στις 24 Απριλίου και στις 26 Ιουνίου με τα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων με αντίστοιχες προτάσεις ε, που θα εξεταστούν εκεί και θα υπάρξει σχετική διαβούλευση. Σας τα λέω όλα αυτά επειδή εδώ πάλι βλέπουμε ναι μεν στο Κοινοβούλιο το μέχρι σήμερα έργο πρέπει να ευχαριστήσουμε για το ότι έγινε και εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά εμείς που βρισκόμαστε εκτός Κοινοβουλίου πρέπει να πούμε ότι στο Συμβούλιο με πολύ έντονο τρόπο και με αντίστοιχη ταχύτητα ή επιτάχυνση προωθούνται αυτά τα θέματα. Πρόκειται εδώ για την άποψη ότι επί της ουσίας διαπραγματεύσεις παράλληλα με τις οικονομικές διαβουλεύσεις θα πρέπει να διεξάγονται. Και σας το λέω ειλικρινά και άμεσα, αυτή την άποψη την ε, συμμερίζομαι διότι ο στόχος πρέπει σίγουρα να είναι ότι φυσικά κατά το τέλος όλων αυτών των διεργασιών ελπίζουμε ότι ο προϋπολογισμός και τα κονδύλια θα εγκριθεί όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκριθούν τα κονδύλια. Είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής δομής ε, για τον προϋπολογισμό, η δομή αυτή να τύχει έγκρισης και παράλληλα λοιπόν με τις οικονομικές διαβουλεύσεις, οι επί της ουσίας συζητήσεις θα πρέπει να διεξαχθούν. Γιατί αν δεν γίνει αυτό υπάρχει ο κίνδυνος, οι πραγματογνώμονες για τα οικονομικά θέματα, τμήματα αυτής της αρχιτεκτονικής δομής να τα αφαιρέσουν και τότε δεν θα είχαμε την δομή αυτή που είχε προβλεφθεί ή θα υπάρξουν τροποποιήσεις που δεν θα ήταν ευκτές. Και υπό το πνεύμα της ε, περιφερειακής πολιτικής που ήταν αντικείμενο των συζητήσεων μέχρι σήμερα είναι σημαντικό τα πιο σημαντικά στοιχεία, τα πιο κέρια στοιχεία αυτής της πολιτικής στην αρχιτεκτονική αυτή δομή, διάρθρωση, να εξακολουθήσουν να υφίστανται, να εξασφαλιστούν. Γι' αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο στη συζήτηση τα πράγματα εκ να προχωρήσουν και να ευδοκιμήσουν. Και γι' αυτό είναι παράκληση που εκφράζω, έτοιμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόσκληση να ακολουθήσουν αυτές τις διεργασίες με αυτό το ρυθμό και με αυτή την τροπή, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο ε, ισότιμα να διαπραγματευτούν, ώστε και οι δύο πλευρές επί της ουσίας ισότιμα από την ίδια αφετηρία να ξεκινήσουν. Και όχι το Κοινοβούλιο να αντιδρά απλώ σε προτάσεις ή τοποθετήσεις του Συμβουλίου. Παράκλησή μου θα ήταν λοιπόν να επιταχύνετε και εσεί το έργο αν γίνεται αλλά πέρα από αυτό φαίνεται ότι προβλέπετε αυτή η επιτάχυνση από πλευρά σας και θέλετε να την ε, προωθήσετε. Αυτά σε σχέση με τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά το Συμβούλιο και τα όσα τεκταίνονται από πλευρά του Συμβουλίου. Είναι κάτι που ήθελα και παρα... Ε, ζητήθηκε από την Πρόεδρο να σας ενημερώσω. Ποια είναι τα κυριότερα σημεία αυτών των πολιτικών. Είναι η σαφής ας το πω έτσι, στοχοθέτηση των επενδυτικών πολιτικών. Μια πολιτική που φυσικά έχει πτυχές υπέρ της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και πρέπει κοινωνικά έτσι να δράσουμε. Επενδύσεις στους ανθρώπους λοιπόν, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις περιφέρειες, ώστε να δημιουργηθεί στο τέλος τέλος πρόσθετη αξία από τις δράσεις μας. Δεύτερο, δεύτερο θεμελιώδες ε, στοιχείο είναι η στοχοθέτηση σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα δεν έχω διακόπτεται ο μιλητής. Δεν έχουμε μεγάλες παρεκκλήσεις ή διαφορές απόψεων. Είναι και σχετικά δύσκολο να διατυπώσει κανείς ενστάσεις κατά του στόχου ότι θέλουμε στο τέλος τέλος όσον αφορά τα χειροπιαστά αποτελέσματα να έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, μετρήσιμα ε, και πραγματικά αξιολογήσιμα αποτελέσματα. Πιο δύσκολο αλλά και πιο ενδιαφέρον είναι το θέμα της συζήτησης που διαμορφώνεται γύρω από τη θεματολογική επικέντρωση ειλικρινά πρέπει να σας πω εδώ ότι δεν ανέμενα και κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον από κάποια κράτη-μέλη που σίγουρα με κάποιες επικρίσεις ή με κροτικό πνεύμα αντιμετωπίζουν προτάσεις. Εκπλησόμεθα όταν ακούμε, ακούμε άτυπα από το Ευρωκοινοβούλιο ότι ο βαθμός εκείνος της θεματολογικής επικέντρωσης τουλάχιστον σε κάποιους τομείς έτσι όπως προτάθηκαν κάποια πράγματα ότι και αυτό ε, μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα και σας το λέω ειλικρινά για τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή και Χέντεγκαρντ. Και δεν είχαν καθόλου εύκολη δουλειά οι συνάδελφοι. Θέλουμε ένα ελάχιστο επίπεδο να διασφαλιστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα στις ενεργειακές επιδόσεις. Έχουν υπάρξει προτάσεις. Είναι μέτρα που, ας το πω έτσι, δεν είναι μόνο για να βελτιωθεί η κατάσταση στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, αλλά και για την διασφάλιση της έδρας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, για την διασφάλιση θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη αν είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτές τις προσπάθειες όσον αφορά τις επενδύσεις και μπορούμε να επενδύσουμε με αυτόν τον τρόπο υπέρ του ανθρώπινου δυναμικού, καλό θα ήταν. Στη συζήτηση θα ήθελα να εξετάσουμε αυτή την πτυχή αυτού του ζητήματος. Θα ήθελα να δούμε κάποια παραδείγματα για σχέδια και προγράμματα για εκείνους τους τομείς και τα παιδεία που δεν καλύπτονται ίσως από τις δικές μας προτάσεις. Διότι πρώτον οι θεματολογικές προτεραιότητες είναι σχετικά ευρείες θα έλεγα. Και όταν έχουμε την προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την πτυχή της καινοτομίας των επιχειρήσεων αυτών και θέλουμε αυτό να προαχθεί, Καινοτομία λοιπόν, όπως το εννοούμε εμείς, όχι μόνο τεχνολογική καινοτομία και νεοτερισμός, αλλά και διοικητικές καινοτομίες και στον τομέα του marketing και στον τομέα των διεργασιών. Όλες οι μορφές και τύποι καινοτομιών και καινοτόμου δράσης καινοτόμων δράσεων που μπορούν να στρέψουν το βλέμμα προς το μέλλον για αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να μπορέσουν η ανταγωνιστικότητά τους να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί. Όλα αυτά είναι στόχοι, στοχοθετήσεις μας και πρέπει όλα αυτά να αντανακλώνται σε μια πολύ πιο αποτελεσματική, ενεργειακά αποδοτική, με εξοικονόμηση ενέργειας πολιτική, οι πολιτικές. Αυτά είναι αυτά που θέλουμε εμείς με τον ένα ή άλλο τρόπο να διασφαλίσουμε να μπορέσουμε να δράσουμε αμφίδρομα. Θα ήθελα λοιπόν επί της ουσίας να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με, παράδει με παραδείγματα όπου θα καταδεικνύεται τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Και αυτό είναι μέρος της διαρθρωτικής πολιτικής σε περίπτωση που δεν καλύπτονται κάποια πράγματα από τις προτάσεις της Επιτροπής. Άλλα θέματα είναι οι όροι και οι, και οι προϋποθέσεις. Εξ άντε, εκ προημίου όροι και προϋποθέσεις. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η αποδοχή ίσως είναι δεδομένη. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που διεξάγονται σε κάποιες χώρες για μια ας το πω έτσι συνταγματική διασφάλιση ή όπου υπάρχει μια ομοσπονδιακή δομή και που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπως από την άλλη πλευρά η Γαλλία όπου οι περιφέρειες με νομοθέτημα, με νόμο δεν επιτρέπεται να έχουν χρέη. Αυτό ε, δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις ε, ε, οικονομικών οριακούς όρου και προϋποθέσεις. Ε, γιατί λοιπόν ε, να ε, κάνουμε κάτι, λένε οι περιφέρειες, που από πλευράς νόμου, νομοθεσίας απαγορεύεται, δηλαδή να συνάπτονται χρέη. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. Οι εκπροημίου προϋποθέσεις και όροι πρέπει στο τέλος τέλος να συνεισφέρουν, ώστε η ποιότητα να αναβαθμίζεται νομοθετικά να μπορεί στο στρατηγικό πλαίσιο να βελτιώνεται, να βελτιώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις δράσης, ώστε τα κονδύλια των διαθροτικών κονδυλίων, τα, των ταμείων, τα κονδύλια να μπορούν ευθύ εξ αρχή να συνεισφέρουν υπέρ αυτών των στόχων. Και φυσικά η γενική ρήτρα Ξέρουμε φυσικά ότι οι, ε, οι δυσκολίες βρίσκονται στις λεπτομέρειες, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και ολοκληρώνοντα κάποια ουσιώδη θέματα όσον αφορά το έγγραφο εργασίας από πλευρά των συντονιστών για την θεματολογική επικέντρωση. Επαρκώς αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα προηγούμενα. Οι μακροοικονομικοί όροι και προϋποθέσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο προανέφερα. Η αρχή τη εταιρική σχέση. Για την εταιρική σχέση πρέπει να πω ότι εξακολουθώ να αναμένω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε εμά σε αυτό το σημαντικό σημείο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά με τα κράτη-μέλη να καταλήξουμε στις συμφωνίες εκείνες που θα συνάψουμε, ώστε με το σωστότερο τρόπο οι περιφέρειες να ενσωματωθούν, να ολοκληρωθούν, να αποτελέσουν μέρος αυτής της ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Και όχι μόνο, αλλά μέσα στην αρχή της πόλη διαχείρισης και πόλη διακυβέρνησης, multi-governance ως θέμα αρχής, να μπορέσουν να δράσουν θετικά. Και θέματα τα οποία συζητώνται εδώ στο τέλος τέλος και που δεν ε, είναι κάτι το απρόσμενο όσον αφορά τις τοποθετήσεις ε, του Κοινοβουλίου και έναντι του Συμβουλίου και η νομική θέση του Common Strategic ε, Framework, του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Αποφασίζεται εδώ η ουσία του εγγράφου αυτός, αυτού και η στοχοθέτησή του θα υποβληθούν σχετικές προτάσεις και νομίζω είναι σημαντικό καταρχήν πρώτα να διασφαλίσουμε την ποιότητα, το υψηλό επίπεδο της συζήτησης και των, και παρεμβάσεων για αυτό το σκοπό. Είναι κάτι το καινοτόμο, κάτι το καινούριο αυτό και για τις υπηρεσίες που πρέπει να αναπτυχθούν, με ποιο τρόπο θα διαμορφωθούν όλα αυτά σε αυτό το πλαίσιο είναι φιλόδοξο και θέτει ίσως και προκλήσεις. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί αυτή η στοχοθέτηση και να δούμε ποιος θα επικεντρωθεί σε ποιο έργο, με ποιο τρόπο. Η κοινή στοχοθέτηση όμως είναι δεδομένη και πρέπει να επιτευχθεί. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ως εγχείρημα. Ιδιαίτερα πολλές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται χρόνο αυτό, δεν το αποκρύπτω. Και για τους αρμόδιους επιτρόπους και τις αρμόδιες επιτρόπους είναι κάτι ως εγχείρημα που ελπίζω ότι θα ευδοκιμήσει με θετικό τρόπο. Ποια νομική συνέχεια θα δοθεί, παραπέρα θα το δείξουν οι συζητήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να αφιερώσω μισό λεπτό για να δούμε πώς θα οργανώσουμε σήμερα ε, τη συνεδρίασή μας, ε, διότι έχουμε μια σειρά παρουσιάσεων και ε, πρότεινα και στους συντονιστές και δεν διαμαρτυρηθήκατε ε, πρότεινα μια κοινή προσέγγιση πρώτα απ' όλα θα έχουμε την εισαγωγή του Ιωάννης Χάν ως εισαγωγή σε όλη τη συζήτηση μετά τη συζήτηση αυτή θα έχουμε ε, από την συνέχεια ε, σε σχέση με την παρουσίασή του και μετά τον Νίκολας Μάρτιν και άλλους ε, για πιο λεπτομερή θέματα. Θα εστιάσουμε ε, το δεύτερο μέρος της συζήτησης στα τέσσερα θέματα για τα οποία ενημερωθήκατε. Θα ήθελα μετά την παρουσίαση του Επιτρόπου να μου επιτρέψετε να ζητήσω από τους εισηγητές και από τους συντονιστές που δεν είναι εισηγητές, διότι υπάρχει μια επικάλυψη ανάμεσα στους εισηγητές και στους συντονιστές όχι πάντοτε βεβαίω, αλλά σήμερα δικαιολογεί αυτή την προσέγγιση και μετά θα περάσουμε σε όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους πρώτους ε, δύο εισηγητές ε, του Γενικού Κανονισμού να λάβουν το λόγο. Παίρνω το λόγο πάρα πολύ ευχαρίστως. Είναι καιρός πια να στρωθούμε στη δουλειά. Έχουμε σημεία στα οποία οι γνώμες μας διαφέρουν. Θα έπρεπε να δούμε <coughs> τι ακριβώς γίνεται, πού βρισκόμαστε. Δεν πρέπει να ξανεφεύρουμε τον τροχό, έχουμε τη στρατηγική 2020, έχουμε τις εκτελεστικές διατάξεις ε, για τη συνοχή, αναφέρθηκαν πολύ σωστά τα διάφορα σημεία. Εμείς ε, προτείναμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, έχουμε μια ομάδα εργασίες ε, για το γενικό κανονισμό και έχουμε και τις εκθέσεις των εισηγητών χωριστά. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα εργαστούμε στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τις πολυετής ε, δημοσιονομικές προπτικές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό φυσικά δεν μας εμποδίζει να στρώθουμε στη δουλειά. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία ή δυνατόν στην πρώτη ανάγνωση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είχαμε πολλές φορές άτυπες συζητήσεις, αναφέρατε δύο ή τρία σημεία, τα οποία εμπλέκουν ε, περαιτέρω διευκρινήσεις την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τα πράγματα μια διαδικασία πιο αναλυτικά, θα γίνει και μία ακρόαση και θα καταθέσουμε μερικές θεμελιώδεις τροπολογίες που θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μαζί και με τις άλλες επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Κάπως έτσι φανταζόμαστε και εμείς την δουλειά μας για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναφέρατε μερικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν ίσως. Αναφέρατε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Μας λέτε ότι πράγματι θα πρέπει να έχουμε διευκρινήσεις να δούμε διαφορετικές προπτικές όπου έχουμε μέσα στη διάθεσή μας τα οποία εφαρμόζονται και υπάρχουν στόχοι οι οποίοι, οι οποίοι ορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο. Μας λέτε υπάρχουν στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στις προτεραιότητες. Θα μπορούσαμε όμως επίσης να δούμε πώς θα τα ενσωματώσουμε όλα αυτά στη διαδικασία συναπόφασης. Ακούσαμε εμείς σήμερα το πρωί το Συμβούλιο το οποίο επίσης βλέπει τα πράγματα μέσα από την ίδια προοπτική. Εδώ και χρόνια ρίχνουμε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον για το τι μπορούμε να κάνουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε. Ας τα ξεκαθαρίσουμε πια τα πράγματα για να μην υπάρχουν πια αμφισημίες. Αναφερθήκατε τώρα στη θεματική συγκέντρωση. Μιλήσατε για ευελιξία και θεματική συγκέντρωση. ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να καταλήξουμε σε άλλους στόχους. Υπάρχουν στόχοι από, για το περιβάλλον, υπάρχουν ε, στόχοι που θα μπορούσαν να καταλήξουν, να αλλάξουν. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε εμείς ποσοστιαίες μονάδες. Μιλήσαμε για το κοινωνικό ταμείο, για την κατανομή αυτό εξαρτάται όμως από το τι παίζεται. Θεωρητικά κάλλιστα μπορούμε εμείς ε, να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο όμως δεν θα ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματικότητα της Βόρειας Φιλανδίας ή της Νότιας Ιταλίας. Χρειάζεται μια σχετική ευελιξία. Θα μπορούσαμε σίγουρα να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε τους θεματικούς στόχους έτσι όπως έχουν διατυπωθεί. Θα ήθελα όμως ευελιξία κατά την εφαρμογή. Εκεί επιμένω πρόκειται για μια ουσιαστική αρχή. Όσον αφορά τώρα στην αιρεσιμότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρίως η μακροαιρεσιμότητα. Εμείς το σκεφτήκαμε πολύ το θέμα. Και ξέρουμε ότι εφαρμόζεται σε χώρες οι οποίες έχουν περιφέρειες ή έχουν μια ομοσπονδιακή διάρθρωση ή στα κράτη-μέλη κάθε αυτά. Όταν έχουμε εμεί το sixth Pack, ξέρουμε ότι έχουμε ένα μακροοικονομικό πρόγραμμα. Έχουμε προγράμματα τα οποία επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει όμως εμείς να βάλουμε προθεσμίες. Όλα αυτά δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα ήθελα όμως να ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένες εξηγήσει για αυτά τα οποία διαμείβονται. Πώς θα λειτουργήσουμε στην πράξη, πώς οι χώρες θα σεβαστούν τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν πριν φτάσουμε δηλαδή στην τελευταία ε, λύση που, στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχει το θέμα του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανατρέψουμε ριζικά τη δομή που φανταστήκαμε. Αυτά ήθελα να πω. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε με κάποιες άλλες συνεδριάσεις που θα μας επιτρέψουν να αναλύσουμε καλύτερα τα πράγματα. Θα έχουμε και την εισήγηση, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά πέστε μας, επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη, ποιες θα είναι οι επόμενες φάσεις. Ευχαριστώ, Νομέρ. Κωνσταντσα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα. Δεν θέλω καθόλου να αναλύσω αυτά τα οποία ανέφερε ο Λάμπερτ Φανίστερ Ροϊ μόλις πριν. Θα έλεγα ότι εντωμεταξύ βρισκόμαστε μέσα στις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις τι θα πούμε σε αυτόν τον κανονισμό, ποιε απόψει και θέσεις θα εκπροσωπήσουμε ω Ευρωκοινοβούλιο και σε κάποιου τομεί ε, εξειδικεύεται ιδιαίτερα αυτό και συμπυκνώνεται ιδιαίτερα. Δεν είναι καθόλου ζήτημα το ότι το Κοινοβούλιο είναι κατά τη συμπύκνωση πόρων και κονδυλίων. Όμως το Κοινοβούλιο, έτσι ερμηνεύω εγώ τη συζήτησή μα, θέλει, θέλει κατά την επιλογή στην οποία θέλουμε να επικεντρωθούμε, να έχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να πούμε ότι θέλουμε να υπάρχουν χρήματα που θα δοθούν στις περιφέρειες και ας κάνουν οι περιφέρειες ό,τι θέλουν με, τα, με αυτά τα κονδύλια. Δεν είναι αυτό το οποίο εννοούμε με ελαστικότητα, εντάξει, όταν προσπαθούμε να υπάρξει ελαστικότητα και ποτέ δεν μου δόθηκε απάντηση σε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι το μέσο, το μέσο το οποίο εσείς πάλι εκ νέου προτείνετε, σε αυτή την εταιρική σχέση συμφωνιών και συμβάσεων εταιρική σχέσης να χρησιμοποιηθεί ίσως με τέτοιο τρόπο ώστε να δούμε την επικέντρωση των ε, κονδυλίων σε συγκεκριμένα θέματα θεματολογικά αλλά και με την αναγκαία ελαστικότητα βέβαια για τις περιφέρειες στην χρήση τους. Γι' αυτό θα χαιρόμουν να πρέπει να πω αν είχαμε πληροφορίες στοιχεία και πληροφορίες για αυτά τα θέματα από το σύμπαν και τον κόσμο εκείνων που ασχολούνται με την πολιτική συνοχή. Είναι αντιφατικά όμως αυτά τα στοιχεία. Ποια μορφή θα πάρουν αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέσης. Θα είναι νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα. Πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά ώστε ναι με τα κράτη-μέλη να είναι ο ένας εταίρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο άλλος συμβαλόμενος εταίρος, όμως οι περιφερειές να εμπλέκονται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι φαντάζεστε σκέφτεστε εσείς, ποιες είναι οι απόψεις σας, τι θα μπορούσε να εξελιχθεί, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η πρόταση. Είναι μια πρόταση που τόσα λίγα, τόσο λίγα αναφέρονται για αυτήν που υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ερμηνεών, ερμηνευτικό περιθώριο. Θα ήθελα με κάποιο τρόπο να τοποθετηθείτε σε σχέση με την πολιτική συνοχή πιο εξειδικευμένα, με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω αν γίνεται στο θέμα της ε, στοχοθέτησης. Εδώ πραγματικά δεν μπορεί κανείς να είναι εναντίον και να έχει διαφωνίες. Ωστόσο, αν αυτές ε, τις προτάσεις ε, δούμε τους δείκτες δείκτες που θα καταλήγουν σε στοχοθέτηση, που θα μετρούν την στοχοθέτηση. Είναι τόσο γενικού χαρακτήρα αυτοί οι δείκτες, σε τόσο γενικό λόγο, γενικό επίπεδο, που θα μπορούσα να πω ότι είμαι υπέρ της ειρήνης, σίγουρα. Είμαι υπέρ της ειρήνης. Κανένας δεν θα διαφωνήσει να είμαστε υπέρ της ειρήνης. Αλλά να δούμε αν σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να έχουμε τέτοιους δείκτες σε ένα τέτοιο κανονισμό. Ή μήπω αν θα έπρεπε με τα κράτη-μέλη άμεσα να διαπραγματευτούμε, να δούμε τι θα ήταν το πιο σκόπιμο να γίνει από πλευρά δικτών, για να έχουμε δείκτε για σωστή στοχοθέτηση γιατί μετά μπορούμε να, κάνουμε, να βάλουμε ένα σημάδι, ένα σταυρό σε αυτά, αλλά δεν θα αλλάξει και τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Σε πολλές συζητήσεις ε, τις τελευταίες εβδομάδες έμαθα κάποια πράγματα τι έμαθα. Δημιουργείται ίσως η εντύπωση στο τέλος τέλος ότι θέλουμε να έχουμε στοχοθέτηση όσον αφορά τα αποτελέσματα, όμως αυτό αντίστροφα πρέπει να σημαίνει ότι θα κάνουμε τους υπολογισμούς με κάθε μολύβι και κάθε χαρτί θα πρέπει να κάνουμε υπολογισμούς προσθέσεις, αφαιρέσεις. Στο τέλος τέλος τα κονδύλια γίνονται όλο και μικρότερα. Πώς θα τα καταφέρουμε, δεν γίνεται αυτό. Θα μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα και για απλούστευση. Αν όλα αυτά τα οποία θέλουμε να εντάσσονται σε αυτές τις προτάσεις συνεισφέρουν στο τέλος τέλος για την απλούστευση. Να έχουμε λιγότερες δαπάνες για ελέγχους για παράδειγμα. Να μην έχουμε τόσο τεράστια έξοδα για δαπάνες και ελέγχους. Γίνονται όλα αυτά καλύπτονται από αυτούς τους κανονισμούς και προτάσεις. Πρέπει από κοινού να στρέψουμε την προσοχή μας πώς μπορούμε να τα πετύχουμε καλύτερα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω αυτό είναι το νόημα εκείνων που αρχίσαμε να συζητούμε στην αρχή και θέλαμε να καθορίσουμε ως τελικό στόχο και να πορευτούμε προς αυτόν, δηλαδή ποια πορεία θα ακολουθούσε η πολιτική συνοχή μας στο μέλλον. Και τα λέω όλα αυτά, λέω ότι το μέσο το εργαλείο του Common Strategic Frames, δηλαδή των κοινών στρατηγικών πλαισίων, θα πρέπει, είναι ενδιαφέρον αυτό, να υπάρξει μια πρόταση στο τραπέζι, να δούμε τι εμπεριέχεται σε αυτή την πρόταση. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συζήτηση επί της ουσίας και θα βρούμε μια οδό, μια πορεία να συμφωνήσουμε προς το συμφέρον όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και στο τέλος τέλος να επιτευχθεί η συμμετοχή, σωστή συμμετοχή, αλλά να υπάρχει και η αναγκαία ελαστικότητα για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές. Νομίζω αυτά είχα να πω. Αυτά είναι κάποια σημεία τα οποία θα έπρεπε να καλυφθούν. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω χωρίς όμως να μπω σε λεπτομέρειες για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Ας φανταστούμε μια κατάσταση όπου θα έχουμε μείωση των κονδυλίων, ότι θα μειωθεί ο προπολογισμό. Ποια θα είναι η αντίδραση και η πρόταση της Κομισιόν. Με ποιο τρόπο θα μειώσουμε την πολιτική συνοχής. Η μείωση των κονδυλίων θα τροποποιήσει το σύστημα ή θα προτείνει άλλες λύσεις η Κομισιόν. Δεύτερον, η γενική φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020. Εμένα μου φάνηκε να κατάλαβα ότι θα είχαμε συνεργαστεί στενά και αποφασιστικά με τα κράτη-μέλη σε επίπεδο προγραμματισμού και μετά θα είχαμε αφήσει ένα μεγάλο περιθώριο ελευθεριών στα κράτη-μέλη για την υλοποίηση στα κράτη-μέλη και θα ελέγχαμε στο τέλος. Δηλαδή, <coughs> θα είχαμε στην αρχή και στο τέλος μία έντονη παρέμβαση, αφήνοντας όμως στη μέση τα πράγματα πιο ήρεμα στη μέση. Τώρα όμως τι βλέπουμε εμείς με την πρόταση που γίνεται, ότι εμένουμε και στο μέσο και υπάρχει και αυτή η μεγάλη θεματολογική συγκέντρωση. Εμείς θα είμαστε υπέρ της συγκέντρωσης όπως είπε και ο κύριος Βανιστερόη και η κυρία Κρέλ. Η ερώτησή μου όπως είναι η εξής. Θέλουμε θεματολογική συγκέντρωση βάσει αυστηρών αρχών ή θέλουμε να υπάρχει μία περιφερειακή τακτοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ποια είναι η αντίληψη που διέπει το όλο οικοδόμημα. Σίγουρα πρέπει να έχουμε αυτή τη θεματική συγκέντρωση, αλλά πρέπει να αφήσουμε και τα κράτη-μέλη ελεύθερα. Στα ADF η θεματολογική συγκέντρωση πηγαίνει ακόμη βαθύτερα. Τι περιμένουμε, πόσο ευρύς πρέπει να είναι ο έλεγχος. Και αυτό αφορά και στις σχέσεις του κανονισμού με των κανονισμών με το CSF. Εμείς έχουμε investment priorities, προτεραιότητες επενδυτικές, που θα πρέπει να καταλάβουμε γύρω από ποιους άξονες κινούνται δεδομένου ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες είναι τόσο συγκεκριμένες. Ρωτώ λοιπόν, είναι λοιπόν τόσο απαραίτητο να μπαίνουμε τόσο πολύ στη λεπτομέρεια και να σταθώ σε αυτό που είπε και η κυρία Κρέλ. Εγώ ως εισηγητής θα προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαγράψει τους δείκτες από τον κανονισμό. ούτως ώστε να τους ξαναδούμε μετά σε μια άλλη νομοθετική πράξη η οποία θα είναι σαφώς αναλυτικότερη διότι θα προσαρμόζει αυτούς τους δείχτες στη συγκεκριμένες πραγματικότητα. Άμα βάλουμε όλους αυτούς τους δείχτες στον κανονισμό, τότε θα έχουμε δείκτες με διαφορετικές παραμέτρους από εκείνες των οικονομολόγων. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και για ποιους δείχτες μιλάμε. Δείχτες απασχόλησης, ε, ποιοι δείχτες θα χρησιμοποιηθούν. Είναι άχρηστο να αναφέρουμε τους δείχτες. Οι δείκτες θα πρέπει να μεταφερθούν σε μια, άλλη, σε μια άλλη νομοθετική πράξη, να μην βρίσκονται μέσα στον κανονισμό. Ξέρω ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα αποτελέσματα, αλλά αν εμείς εδώ πάρουμε τους δείκτες και τους γενικεύσουμε στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, θα έχουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει νόημα. Και μια άλλη ερώτηση για τον κώδικα συμπεριφοράς και τις ε, ε, συμβάσεις, τις ε, συμφωνίες συνεργασίας. Θα υπάρχει κώδικας συμπεριφοράς ε, για τις ε, συμφωνίες συνεργασίας, ε, τον οποίο θα φτιάξετε εσείς ή θα το αφήσετε στα κράτη-μέλη. Τελευταίο λοιπόν, προς τα που τίνουμε, προς την ευελιξία ή προς την αυστηρότητα και τον προκαθορισμό. Ήθελα επίσης να πω συναδέλφους ότι θα συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται ο Επίτροπος να μπει σε λεπτομέρειες για κάθε θέμα, να μας δώσει τις πολιτικές ε, γραμμές. Έχετε το λόγο. No, uh, Πρώτα απ' όλα, σχετικά ε, μίλησα για το θέμα ε, της νομικές θέσεις του CSF είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε αργότερα. Για την ώρα είναι πιο σημαντικό να έχουμε μια κατάλληλη πρόταση να συζητήσουμε το περιεχόμενο και ίσως θα υπάρξει μετά τελικά το, το, το, νομικό καθεστώς του CSF. Νομίζω ότι θα πρέπει για την ώρα να έχουμε μια καλή πρόταση για αυτό το νέο θέμα. Σχετικά με τους μακροοικονομικούς όρους, βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ίσως μια χωριστή συζήτηση για ποια είναι η κοινή γνώμη της Επιτροπής. Έχουμε με την ΕΚΟΦΗΝ και με άλλους ε, συζητήσεις πώς παρουσιάζονται θεωρητικά τα πράγματα, διότι είναι ένα μέτρο ε, τελευταίας καταφυγής που θα πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να συζητηθεί, να δούμε ποιες είναι οι ιδέες. Ε, θα μπορούσα να επανέλθω όχι, με, όχι με την ιδέα, αλλά για να συζητηθεί εδώ. Ξέρω, ξέρω. Δεν είστε οι μόνοι που το σκέφτεστε αυτό σχετικά ε, με την ποιότητα των συμβάσεων εταιρική σχέσης. Ε, πρόκειται για μια ε, συμφωνία που καλύπτει πολλά πράγματα, μια ομπρέλα που καλύπτει πάρα πολλά πράγματα, αποτελέσματα που συμφωνήσαμε και βεβαίως εξαρτάται αυτό από το νομικό πλαίσιο μιας χώρας, ενός κράτους μέλους. Ποια είναι η πολιτική ποιότητα εφαρμογής ε, Λαμβάνοντα υπόψη την περιφέρεια που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Λόγω της πολυεπίπεδης προσέγγισης θέλουμε περιφέρειες αλλά και τοπικές αρχές που να εμπλακούν πολύ περισσότερο στις διαπραγματεύσεις. Αλλά τελικά αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, αλλά όπως είπα και συχνά εδώ, πιστεύω ότι ήδη η ε, δημιουργία αυτού του άρθρου στον κανονισμό είναι, αν θέλω, μια, ένας πολιτικός ισχυρισμός αρκετά ισχυρός για το τι πρέπει να γίνει. Σχετικά με τους δείκτες, πρώτα απ' όλα, αλλά ίσως αυτό να μπορεί να συζητηθεί αργότερα με τον Νίκολας Μάρτιν, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους δείκτες ε, αποτελεσμάτων ε, και τα αποτελέσματα. Ε, οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι τα, είναι τα χιλιόμετρα οδών που κατασκευάζονται. Και είναι σαφές ποιος πρέπει να είναι εκεί ο τελικός στόχος. Πρέπει να πω και ε, και υπήρξαν συζητήσει στην αντίστοιχη ε, ομάδα εργασία και η πρόκληση ήταν να βρεθούν κοινοί δείκτε που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ε, σε όλε τι 27 και αργότερα 28 χώρε μέλη. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και ορισμοί για την ίδια έννοια σε πολλές χώρες. Βασιστήκαμε πολύ στην Eurostat σχετικά με τον ορισμό των δικτών και χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, ο κατάλογος των δυνητικών δικτών δεν ήταν τόσο μακρύς. Υπάρχει μια πρόταση, υπάρχουν συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε που έχει οριστεί αυτό, που έχει προσδιοριστεί και θα είναι θέμα περαιτέρω συζητήσεων για την ώρα. Πρέπει να βρούμε μια συμφωνία για το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτών των δικτών. Απλούστευση και πάλι θα πρέπει να είναι κάτι που χρειάζεται μια ολόκληρη συνάντηση για να συζητηθεί και να έχουμε εμπειρογνώμανες με τις γνώσεις τους. Θα μπορούσα να ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να μας δώσουν ένα κατάλογο, μια σύνθεση για τη διάρκεια, για την διάρκεια όταν έχουμε ένα αίτημα πληρωμής, μια απέτηση, πόσο χρόνο χρειάζεται μέχρι ο τελικός δικαιούχος να πληρωθεί. Κατά τη διάρκεια των αποστολών μου έχω διαπιστώσει ότι καμιά φορά χρειάζεται και η μεγαλύτερη διάρκεια ήταν δύο χρόνια. Σε άλλη χώρα οκτώ μήνες, ε, μέσα στο επίπεδο της Επιτροπής είναι ένας έως δύο μήνες. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στους άλλους 22-23 ε, μήνες. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος, de facto. Υπάρχει πολλή κολλησιεργία στα κράτη-μέλη και ε, τα κράτη-μέλη ξέρουν ότι η έγκριση ενός έργου απαιτεί καμιά φορά 63 υπογραφές στο φάκελο. Κάποιος έλεγε με κοινικό τρόπο ότι αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν υπογράψει αυτήν την ένταση έχουν 1,6% ευθύνη. Δεν είναι αυτή η κατάλληλη προσέγγιση. Ας συζητήσουμε μαζί για την απλούστευση. Ε, μπορώ να πω ότι και στόχος μας είναι να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στις περιφέρειες, στις χώρες όπου έχουμε γνώση αποδείξεις ότι όλα λειτουργούν καλά και γνωρίζουμε τους πελάτες μας και αυτό σημαίνει ότι κυρίως όσον αφορά στις δραστηριότητες ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, σημαίνει διαφοροποίηση στο μέλλον σχετικά με την επένδυση σε ανθρώπινους πόρους. Αλλά επίσης ως ό,τι αφορά την συνέχιση των θεμάτων συμμόρφωσης, αν πρέπει να επαναληφθεί όλη η διαδικασία σε μια χώρα όπου με τη σημερινή προοπτική όλα πηγαίνουν καλά, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί ολόκληρη η ιστορία και είναι ευκολότερο να συνεχίσουμε. επανερχόμενος στην θεματική συγκέντρωση. Αναφέρομαι στην πρότασή μας, ίσως την επαναλάβω. Εάν μιλήσουμε μόνο για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουμε προτείνει για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις, τον νέο τύπο των μεταβατικών περιφερειών, Ξέρετε ότι στις περιφέρειες αυτές τα διαθέσιμα κονδύλια σε σύγκριση με τα λιγότερες ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι επίπεδα αρκετά χαμηλά. Γι' αυτό προτείναμε συγκέντρωση των διαθεσίμων πόρων και η πρότασή μας ήταν και είναι ότι 80% των διαθεσίμων ε, κονδυλίων ε, για μια δεδομένη περιφέρεια θα πρέπει να ξοδεύεται για τρεις στόχους. Πρώτον, καινοτομία, έρευνα, ανάπτυξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και μετά ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες, ε, τουλάχιστον 90% από αυτά, τα 80% θα έπρεπε να διοχετεύεται προς την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και σας ρωτάω, με τις τρεις, τρεις αυτούς στόχους, έχετε ακόμη 20% ε, χρήματα που δεν έχουν προσδιοριστεί. Ποιοι είναι οι τομείς όπου δεν βλέπετε την δυνατότητα να έχετε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα. Και για το 20%, 5% για την ανάπτυξη αστικών κέντρων και πόλεων. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει καθορίσει αυτό για την αηφόρο ανάπτυξη των κέντρων. Νομίζω ότι στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες έχουμε μια κατάσταση που θα συνεχιστεί στο μέλλον, όπου δεν χρηματοδοτούμε υποδομές. Γι' αυτό για τις ολιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες έχουμε μόνο 50% ε, διάθεση για αυτούς τους τρεις στόχους. Ναι, υπάρχει 5% όπως είπατε ε, για τη διάθεση για τις αστικές περιοχές, αλλά νομίζω ότι περισσότερες επενδύσεις στις αστικές περιοχές είναι για την ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, μόνωση κλπ. Είναι ένα άλλο παράδειγμα, ένα καλό παράδειγμα του πώς όλες οι ιδέες ε, που πλανώνται γύρω μας μπορούν να ενταχθούν στις προτεραιότητές μας. Και έχουμε υπολογίσει εκ νέου για, με τις τρέχουσες πρόπτικες. Νομίζω 92-93% όλων των κονδυλίων που πραγματικά ξοδεύονται μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις προτεραιότητες. Μετά έχουμε την πολιτιστική κληρονομιά κλπ. Και αυτό θα είναι εφικτό στο μέλλον το μόνο πράγμα είναι οι περιφέρειες. Σύμφωνα με τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν ποια, πώς θα εστιάσουν ορισμένες επενδύσεις. Ε, μέσα σε αυτό το αρκετά ευρύ πλαίσιο και αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που λέμε εστίαση και προσαρμογή στην πραγματικότητα, συγκέντρωση ε, και λύσεις κατά παραγγελία. Νομίζω ότι όλα τα κρατημέλη και οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αναπτύξουν λύσεις κατά παραγγελία προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους ε, και στα αιτήματά τους, στις απαιτήσει τους. Αυτό που είπε ο Γιάνν Όλμπριχτ για τον προϋπολογισμό αυτό εξαρτάται για την ώρα. Η υπόθεσή μας είναι να πάρουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε ζητήσει. Αλλά γι' αυτό έχω ήδη πει στην εισαγωγή μου ότι θα εκτιμούσα και θα πρότεινα πραγματικά να διαπραγματευτούμε το περιεχόμενο παράλληλα με την χρηματοοικονομική διάσταση. Διότι αν συζητηθεί πρώτα ο προϋπολογισμός και τα οικονομικά θα υπάρξει ε, κίνδυνος ε, μερικά κομμάτια να αποσυρθούν. Και ξέρετε ότι ένας από τους στόχους είναι πάντοτε η εδαφική συνεργασία. Ένας άλλος μπορεί να είναι οι μεταβατικές περιφέρειες όπου οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλότερες και να δούμε το μερίδιο αυτών των νέων μεταβατικών περιφερειών. Πρέπει να έχουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις παράλληλα ε, για να αποφύγουμε ε, να πληγεί όλη η αρχιτεκτονική. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν παράλληλα αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εάν τελικά υπάρχει μία μείωση, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω ήδη να μιλάω για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά θα πρέπει τότε να δούμε τα πράγματα γραμμικά και να μην αφαιρέσουμε το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα σημείο πολύ ενδιαφέρον, πάνω στο οποίο θα ήθελα να επισύρω την προσοχή του Κοινοβουλίου. Έχουμε, την, θα έχουμε τους νέους πίνακες σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ και θα νομίζω ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση του ΑΕΠ και αν υπάρχει πάντοτε μια συζήτηση με 1%, κάτι λιγότερο από 1%, κάτι λίγο περισσότερο από 1%. Κάποια στιγμή θα κρυθεί απαραίτητο ε, να μιλούμε με απόλυτους αριθμούς, διότι εάν υπάρξει σημαντική μείωση του ΑΕΠ 1% ή ε, κάτι λιγότερο από 1%, αυτό θα είναι χαμηλότερο από ό,τι φαντάζεται κάποιος για την ώρα. Γι' αυτό ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε αυτό το θέμα που θα βρεθεί επιτάπητο σε μερικές εβδομάδες το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Θα λάβουμε τα τελευταία στοιχεία τότε. Σχετικά με την εδαφική υπευθυνότητα, συμμερίζομαι την προσέγγιση σας, πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός, αν σας κατάλαβα καλά, ανάμεσα στις περιφέρειες και τα κρατη και να δούμε ποιος κάνει τι Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 25 λεπτά έχουμε. 14 αγορητές. Δεν θα τα καταφέρουμε με αυτή την ταχύτητα να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Ζήτω από τους τέσσερις ε, εισηγητές ε, που απομένουν να είναι το δυνατόν πιο σύντομοι. Στενάρου, ε, Φέιον και Μαρία στη συνέχεια η Ριγκόεν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, επειδή πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ κάπως και πιο συγκεκριμένα σε ένα ρουμανικό θέμα. Θα μιλήσω ρουμανικά λοιπόν. Φορέστε τα ακουστικά σας. Ήθελα να πω ότι την Δευτέρα στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, στο, στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργός ε, ε, ξεκίνησε ασύστατες και αδικαιολόγητες επιθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ε, η αντιπολίτευση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και η Σοσιαλφιλελεύθερη Ομάδα ζήτησαν λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει την χρηματοδότηση με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ρουμανίας. Απέστειλα μια επιστολή εχθές προς τον Επίτροπο Χάν και σήμερα το πρωί πήρα μια πολύ θα έλεγα πολιτισμένη απάντηση που αρνείτο τέτοιου είδου ε, κατηγορίες και χρησιμοποιώ την ευκαιρία, δράτω με αυτής της ευκαιρίας, να ευχαριστήσω προσωπικά τον Επίτροπο Χάν. Σα τιμά αυτή η απάντηση, Επίτροπε Χάν, και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι όπως απαντήσατε. Η ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη, η ευρωπαϊκή ατζέντα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής. Ακόμα και στη Ρουμανία που αντιμετωπίζει πραγματικά θέματα απορρόφησης κονδυλίων. Και για το μέσο της διευκόλυνσης Europe Facility. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για μια τέτοια κατάσταση, όπου όχι μόνο οι βουλευτές, αλλά και στο Συμβούλιο βλέπουμε ότι υπάρχει επίμαχο θέμα για τον, τρέμα, με τον τρόπο με τον οποίο δέκα δισεκατομμύρια θα αφαιρεθούν από το Ταμείο Συνοχής για να μπορέσουν να διατεθούν στο Ταμείο Διευκόλυνσης, στη διευκόλυνση ως μέσο. Δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες, αποκεντρωμένη διαχείριση, κεντρο, κεντρική κτλ. Μέχρι σε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα μια σαφή απάντηση. Γιατί, πώς, ποιες είναι οι αρχές, ποια είναι τα κριτήρια Πώς θα μετρηθούν τα ωφέλη και τα θετικά αποτελέσματα. Δώστε μας πρώτα, Επίτροπε, λόγους για να δεχθούμε αυτή την πρόταση ως ιδέα και μετά δεύτερο στη συνέχεια να δούμε αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ή όχι. Και για τα θέματα ενέργειας και από τη δική σας δήλωση εγώ μπορώ να συναγάγω το συμπέρασμα ότι είναι ζωτική σημασία ακόμα και το Ταμείο Συνοχή ε, να μπορέσει να αποτελέσει πεδίο άντληση κονδυλίων ε, για αυτέ τι δράσει λόγω των κοινωνικών επιπτώσεων είχα επαφή με δύο επιτρόπους και ε, ήμουν σε επαφή και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Όλοι είναι υπέρ της ε, διασφάλισης ε, όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής για τα θέματα στέγασης, θέρμανσης κτλ. Θα ήμουν ευγνώμων αν και εσείς προσθέτατε τη φωνή σας σε αυτή τη στάση που είναι θεμελιώδου σημασία για την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης κονδυλίων. Τέλος, πώς θα συνεργαστείτε με τον Επίτροπο Ποτόσνικ για να διασφαλίσετε ότι οι νέες οδηγίες ε, μελέτης αξιολογικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, επιπτώσεις εξέτασης ε, των, ε, συνεπειών στο περιβάλλον <clears throat> δεν θα αλλάξουν ή θα τροποποιηθούν κατά κάποιο τρόπο διότι από το άρθρο 177 της συνθήκης και το 100 ε, εδάφιο 5 αναφέρεται ότι μόνο στην περίπτωση που ο ρηπαντής, ο ρηπαίνων δεν πληρώνει, τότε το Ταμείο θα πρέπει να αναλάβει τα κόστη της ε, μεγάλης ε, εμβέλειας ρήπανσης ή μόλυνσης. Εμείς όμως θέλουμε να πούμε ότι είναι θέμα έσχατης προσφυγής, εξτρέμα ράτσιο και όχι κάτι το συνηθισμένο κάτι το ξεχωριστό δηλαδή και κατ' και όχι κάτι το συνηθισμένο. Να συνεργαστείτε με τον κύριο Ποτόσνικ παρακαλώ να διευρυνθεί το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προληφθεί, να αποφευθεί η, η ε, πιθανότητα αυτή να δημιουργηθούν τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις δηλαδή αντί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σας ευχαριστώ. Ρίκα, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια εξαιρετική παρουσίαση από πλευράς της. Ουσιαστικά θα ήθελα κάποια σχόλια να κάνω σε σχέση με τα θέματα που καλύφθηκαν εν συντομία. Θεματική επικέντρωση, θεματολογική επικέντρωση, όπως προανέφεραν και άλλοι βουλευτές. Μπορούμε ω Κοινοβούλιο να υποστηρίξουμε μια τέτοια προσέγγιση, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα τον κανονισμό ETC, ε, ε όπου έχω αναλάβει εγώ την εισήγηση, δεν ταιριάζει με ένα τέτοιο τρόπο στο ETC ε αυτή η πρόταση και στους στόχους του ETC. Πολλά θέματα αγνοήθηκαν ξέχασαν να τα καλύψουν. Ιδιαίτερα την προώθηση και την προαγωγή της ε, διαμεθοριακής συνεργασίας. Θέματα για παράδειγμα επίσης και των μεταφορών. Θέματα μεταφορών που απουσιάζουν επίσης. Θα πρέπει να δούμε τα θέματα του ETC. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και θα πρέπει περισσότερα να επιλεχθούν από τους τέσσερις άξονες που αναφέρονται, τα τέσσερα θεματικά πεδία που αναφέρονται και να προκαθορίζονται κονδύλια προς τη χρήση τους, earmarking. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε κάποιες χώρες ε, αυτό ίσως μπορεί να δημιουργεί κάποια προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαφορετική αφετηρία ως σημείο για θέματα περιβαλλοντικά των διαφορετικών κρατών. Θα ήθελα λοιπόν με περισσότερο κριτική κριτική φωνή και κριτικό πνεύμα να αντιμετωπίσω αυτή την πρόταση. Τώρα, όσον αφορά αυτού του είδους τις συμβάσεις και συμφωνίες που μπορούν να βοηθήσουν και αυτό θα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτή την πρόταση στο κείμενο και μάλιστα και με δεσμευτικό χαρακτήρα. Σε κάποιες χώρες υπάρχει μεγάλη ανησυχία οι περιφέρειες να μην βρεθούν εκτός ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων και, και αυτές να μπορούν να συμμετέχουν δηλαδή ισότιμα με άλλα λόγια. Θα ήθελα στον κανονισμό ETC να δούμε πόσο πραγματιστικά μπορεί να συνδεθεί με συμβάσεις και συμφωνίες εταιρικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τους δείκτες, ένα επόμενο σημείο. Θα ήθελα πραγματικά να μου δίνατε κάποιες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες εξειδικευμένες ε, παρατηρήσεις να κάνετε και όσον αφορά και την περιφερειακή ε, συνεργασία θα, καλό θα ήταν ε, από πλευράς εγγράφων να έχουμε μια ε, ας το πω έτσι, πιο ξεχωριστή τοποθέτηση σε σχέση με τον κανονισμό και για την απλούστευση. Και για την απλούστευση θα θέλουμε να έχουμε σαφέστερες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή την περίοδο προγραμματισμού έχουμε θέματα απλούστευσης όπως κατά ποσά ε, ποσά τα οποία υπολογίζονται και καταβάλλονται ε, διαμιάς ε, ή προκαταβολές. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά και για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και την προσέγγιση αυτή. Διερωτώ με σε ποιο βαθμό και πώς θα καθοριστούν τα προγράμματα στην πρακτική εφαρμογή από αυτές τις αρχές και ποιο θα είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών και συμβάσεων εταιρικού χαρακτήρα, εταιρική σχέση. Είναι λοιπόν σημαντικό όχι μόνο να επικεντρωθούμε και να ασχοληθούμε με το πλαίσιο, πρέπει να είναι τα κατόφλια πιο εύκολο να επιτευχθούν, να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, προσπελασιμότητα στο εφικτό της προσπάθειας. Και μετά όσον αφορά της, ε, τη μεταβατική περίοδο, τη μεταβατική κατηγορία, θα ήθελα να υποβληθούν αριθμητικά μεγέθη συγκεκριμένα για το τι θα σήμαινε αυτό για αυτές τις κατηγορίες. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι αν οι περιοχές σύγκλησης μεταφερθούν, μετατραπούν με αυτόν τον τρόπο σε διάμεσες περιφέρειες, ε, ενδιάμεσες κατηγορίες, ο πληθυσμός ε, θα συρρυκνωθεί, δηλαδή, θα είναι μικρότερος ο αριθμός των ατόμων που θα υποφεληθούν σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες. Και στην μεταβατική κατηγορία τι θα γίνει στις μεταβατικές κατηγορίες. Με το phasing in, phasing out, άλλες κατηγορίες θα αυξηθούν πληθυσμιακά. Πρέπει να δούμε αυτές τις διαφορές Καταρχήν το κόστος θα αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά αν συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με εκείνη που θα δημιουργηθεί στο μέλλον με το νέο προγραμματισμό και τις νέες ενδιάμεσες κατηγορίες με αυτές τις μεταβατικές κατηγο... ενδιάμεσες κατηγορίες μπορείτε να αποσαφηνίσετε αυτή την ερώτηση τι θα σημαίνουν όλα αυτά σε αριθμητικά μεγέθη με τις νέες κατηγορίες και με τα κόστη αν δημιουργηθούν αυτές οι ενδιάμεσες κατηγορίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Χάν, Ευχαριστώ για το ότι μπορούμε και πάλι να ξανασυζητήσουμε μαζί σας. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονική τομή αυτή ως χρονικό σταυροδρόμι. Ιδιαίτερα και όσον αφορά και το ε, θέμα για το οποίο είμαι εισηγητής ε, θα είχα πολλές επιμέρους ερωτήσεις. Μπορώ όμως ε, και με τους διευθυντές υπηρεσιών σας και με τους υπεύθυνους συνεργάτες σας να διευκρινίσω αυτά τα θέματα. Αυτό το οποίο με κινεί περισσότερο ως μέλημα είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Πώς εσείς ως υπεύθυνο επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική θα αντιμετωπίσετε την αντιπαράθεση που διεξάγεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι των συναδέλφων σας, αλλά και στο Συμβούλιο σε σχέση με τις συζητήσει που βρίσκονται υπό εξέλιξη και όχι μόνο αφορούν τους πολίτες αλλά και τις κυβερνήσεις παράδειγμα υπό την έννοια χρέωση, ε, υπερβολικό χρέος, οικονομική σταθεροποίηση, προγράμματα σταθερότητας και λιτότητας και ο τύπος βρήθη από κρίσεις για μείωση και ύφεση των οικονομικών επιδόσεων, ύφεση στην οικονομία και προβλέπονται προβλέπεται αύξηση του αριθμού των ανέργων στην Ευρώπη λόγω αυτής της ύφεση και συρρήκνωσης οικονομικής και έχουμε και προτάσεις ε, για το, κοινωνικό, για το στρατηγικό, κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τις πολιτικές συνοχής και στήριξης. Βλέπω όμως ότι από τους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε ένας βλέπει μόνο τα δικά του συμφέροντα, του δικού του τομέα. Εκεί όπου έχουμε κομβικά σημεία που συνδέουν τις επιμέρους πολιτικές με άλλες, αγνοούνται τα πράγματα. Εκεί που πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κοινή δεν δίνεται σημασία σε αυτά τα κομβικά σημεία. Τι είναι η περιφερειακή πολιτική και τι είναι ο ορίζοντα, χρονορίζοντας 2020. 2020. Ποια είναι τα αποτελέσματα συνέργεια και οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής συνέργεια και δράσης. Βλέπετε υπάρχουν πολλά ερωτήματα και υπογραμμίζουν τις αβεβαιότητες και ανασφάλειες που αισθάνονται και οι συνάδελφοι όπως εκφράζονται στις παρεμβάσεις τους. Έχουμε, είχαμε και την Πολωνική Προεδρία προηγούμενα που με καλό τρόπο και με θετικό τρόπο τέθηκε στα θέματα και υπέρ του ιδίου συμφέροντος για την διαφορετική πολιτική και την ε, πολιτική ε, της σύγκλησης και συνοχής. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση του δανέζικου προγράμματος της Προεδρίας από τον Δανό, Δανέζο Υπουργό. Ρωτήθηκε κατά πόσο θα συνεχίσει το πρόγραμμα της Πολωνίας και είπε, ας το πω ευγενικά αυτό το οποίο ανέφερε, ήταν επιφυλακτικός τουλάχιστον επιφυλακτικός και για τα θέματα της πολιτικής συνοχής θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα ώστε η Δανέζικη Προεδρία να μπορέσει να δράσει όπως ε, θα έπρεπε και θα, μέχρι, μέχρι δύο ημερομηνίες που προανέφερε, όπου η Δανέζικη Προεδρία στοχεύει να εγγράψει αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη τον Απρίλιο, λέει, και τον Ιούνιο, με δύο μεγάλες, μεγάλες συνόδους. Ε, μέχρι τότε τι θα γίνει ε, θα έχουμε λέει είπε άτυπε συζητήσει σε Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει προγραμματιστεί κάτι άλλο, τίποτα άλλο δεν προβλέπεται. Σε μια χρονική στιγμή όπου ακριβώς τα θέματα επί τη ουσία, όπως ε, έχουν τεθεί εδώ ενώπιό σα πρέπει να αποσαφινιστούν άμεσα για να δράσουμε αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν αμφιβάλλουμε όσον αφορά τα θέματα της μακροοικονομικής ε, πολιτικής όρους και προϋποθέσεις που τίθενται που αν θα έπρεπε να είναι ή όχι αντικείμενο της πολιτικής συνοχής. Όμως ο συνάδελφος Μποστινάρου τι είπε. Είπε ότι το ρουμανικό παράδειγμα, και το διαβάζουμε αυτό σήμερα στα δημοσιεύματα στις εφημερίδες, απειλήθηκε λέει η Ουγγρική κυβέρνηση, η Ουγγαρία, ότι αν δεν προσαρμοστεί σε σχέση με τις ε, συστάσεις που έγιναν Δηλαδή, μια πρακτική που ακολουθείτε, που αποκτά ε, σάρκα και οστά με τέτοιου είδους ε, συστάσεις και πολιτικές που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα λοιπόν, διατυπώνετε το ερώτημα, πώς εσείς τοποθετήσετε σε τέτοιου είδους προκλήσεις, ποια είναι τα επόμενα βήματά σας και διαβήματα για να διασφαλίσετε τι θα γίνει με την πολιτική συνοχή και τη διαφορετική πολιτική, ώστε επιτέλου να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν οι περιφέρειες τη Ευρώπη και να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. Και για να μην είναι μέσο ή εργαλείο ίδια συμφέροντα, ιδιωτελώ ε, συμφεροντολογικά να προωθούνται και μόνο έτσι να ε, τίθενται στο προσκήνιο για να επιτευχθούν άλλοι πολιτικοί στόχοι αγνοώντας την ουσία ή θέτοντας στο κέντρο βάρους εκεί όπου εξυπηρετούνται κάποιοι να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς δηλαδή τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ. Η θετοντας το κεντρο Ιριγκόγεν. Ελπίζω να είσαστε πιο σύντομοι εσείς κυρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Κύριε πίτροπε λυπάμαι αλλά όλοι θα πάμε προς την ίδια κατεύθυνση, στον ίδιο, τον ίδιο δρόμο θα πάρουμε σε αυτή την Επιτροπή, γιατί συμμερίζομαστε όλοι τα ίδια κριτήρια. Και εγώ ως εισηγήτρια της γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα συγκεντρωθώ στα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Θεωρώ ως εισηγήτρια πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το 25% του κοινωνικού ταμείου στους καιρούς που περνάμε. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε σταθερό το ταμείο, πρέπει να αποτελεί κλειδί για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει όμως και η απασχόληση που θα δημιουργηθεί να είναι αηφόρα, να είναι διαρκής για να μπορέσει να απορροφήσει αυτούς που είναι άνεργοι καιρό. Θα πρέπει να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και τους υψηλούς δείχτες φτώχειας. Για τα ελάχιστα ποσοστά που μιλάμε, 25, 40 και 52, η πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα στη χρήση των κονδυλίων και η απορρόφησή τους. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να επιβάλλουμε σταθερό ποσοστό για κάθε περιφέρεια διότι όλες οι περιφέρειες δεν είναι κομμένες με το ίδιο πατρόν. Επίσης, θεματολογική συγκέντρωση και ευελιξία. Φυσικά πρέπει να είμαστε συνεπείς με τη στρατηγική 2020. Αλλά πολλές φορές είπαμε στον Επίτροπο ότι η πολιτική συνοχή είναι κάτι παραπάνω από ότι ένα μέσο της στρατηγικής 2020. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ενσωματώσουμε και μία ευελιξία για να λάβουμε υπόψη μας τις ειδικέ ανάγκες της κάθε περιοχής, να δούμε την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της στόχιας. Έχουμε επίσης 18 προτεραιότητες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι με αυτές και στη χρηματοδότησή τους, διότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις ανομαλίες που θα δημιουργούσε ένα ενιαίο καλούπι για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες οι οποίες δεν είναι όλες ίδιες. Στην πρόταση της Κομισιόν αυτό δεν είναι σαφές. Πρέπει να ορίσουμε τον ρόλο των όσων συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Πρέπει να φύγει σε 10 λεπτά ο Επίτροπος και έχω σας παρακαλώ, ναι, αν θέλουν οι συντονιστές να θέσουν ερωτήσεις, ας το κάνουν, αλλά για τη συζήτηση θα το κάνουμε μετά όταν θα έχουμε τον Νίκολας Μάρτιν μαζί μας. Μόνο για αυτούς που θέλουν, ε, Νέσκο, ο Μαντζή, αν έχετε ερωτήσεις, μόνο ερωτήσεις. Έχω ένα μακρύ κατάλογο για μετά. Όποιος θέλει να θέσει ερώτηση από τους συντονιστές Ραμόνο Μανέσκου. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη λόγω της πίεσης χρόνου. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, μέχρι ποιου βαθμού μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι με τη ε, θέση σας ε, στο Κολέγιο των Επιτρόπων θα μπορέσετε να υπερασπιστείτε την πολιτική ε, της συνοχής όσον αφορά την μακροαιρεσιμότητα για να αποφύγουμε κατάσταση όπου η πολιτική συνοχής θα γινόταν το βασικό μέσο για κυρώσεις σε κράτη που δεν ε, έχουν καλή επίδοση. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα κάνετε κάτι για την απλούστευση. Έγινε πάρα πολλής λόγος για την απλούστευση, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία διότι δεν είναι αποτελεσματικό να ε, επιβάλλουμε το ίδιο ποσοστό στα κράτη-μέλη χωρίς να παίρνουμε υπόψη ε, το, το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιφέρειας, κάθε χώρας και τις ανάγκες. Έχουμε και την αστική ατζέντα. Θα μπορούσαμε ίσως να αναθεωρήσουμε αυτό τον κατάλογο των 20 πόλεων και οι κοινοί δείκτες που αναφέρθηκαν ευνοούν τις μεγάλες πόλεις, αλλά δεν απαντούν ε, στις ανάγκες αστικής ανάπτυξης των κρατών μελών. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ο περιορισμός της χρηματοδότησης που παρέχεται σε μεγάλες εταιρείες. Λόγω της προηγουμένης περίοδου είδαμε ότι υπήρχε καλή συνεργασία ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να διαφυλάξουμε την δυνατότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ε, ούτω ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις να μπορούν να δικαιούνται και να υποφελούνται ε, από χρηματοδότηση σε συνεργασία με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι θέλουμε να τις υποστηρίξουμε. Κύριε Επίτροπε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να καλύψω αυτό που ζήτησε η Πρόεδρος. Το στρατηγικό πλαίσιο είναι και το γερό κομμάτι της όλης σας πρότασης. Θα θέλαμε όμως να είναι πιο ορισμένο. Και έτσι εμείς θα μπορούσαμε να άρουμε μία αμφισημία. Η πολιτική συνοχής δεν είναι στρατηγική 2020. Συμπεριλαμβάνει στόχους τη στρατηγική 2020, αλλά δεν είναι η στρατηγική 2020. Είναι κάτι που πάει πολύ πιο μακριά, βρίσκεται μέσα στη συνθήκη. Εσείς είστε πολύ περιορισμένος στη στρατηγική 2020. Ένα ειδικό επίσης πρόβλημα για μας είναι το θέμα του σπασίματος της συνοχής Μπορεί να έχουμε σε μία περιοχή προβλήματα περιβάλλοντος, αλλού δημογραφικά προβλήματα, άλλη περιφέρεια η οποία να πλήττεται από μία τεράστια οικονομική κρίση και να έχει προβλήματα απασχόλησης. Θα έπρεπε λοιπόν η κάθε περιφέρεια να μπορεί να συμμετέχει στο διάλογο με την Κομισιόν και να συνεισφέρει στο πρόγραμμα που ορίζεται για αυτήν. Επίσης, τα διαρθρωτικά προγράμματα που αναφέρετε εσείς και που αποτελούν ένα σπάσιμο της συνεχής, μιλάτε για το 174 άρθρο της Λισαβόνας και κάνετε μία διάκριση μεταξύ των αρεοκατοικημένων περιοχών, τις ξεχωρίζετε από τα νησιά, ε, δεν τις ξεχωρίζετε από τα βουνά. Πώς θα μπορούσαμε όμως εμείς να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο μεταξύ Φεντέρ και Φεαντέρ το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στην ε, πρότασή σας. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάνω, παραπάνω στοιχεία. Αυτό για τις ενδιάμεσες περιοχές τις υποστηρίζουμε. Πρόκειται για κάτι το καινούριο στην πολιτική συνοχής. Το σχέδιό σας τη συμπεριλαμβάνει πολύ καλά για τα κονδύλια που τους δίνονται και τη συγχρηματοδότηση, αλλά όχι για την ευελιξία. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει και μία ενδιάμεση ευελιξία. Και τελευταίο σημείο που κανένας δεν αναφέρθηκε είναι η απλούστευση. Διαβάζοντας το κείμενό σας, διαπιστώνουμε ότι η απλούστευση εφαρμόζεται για να κάνει τη ζωή πιο εύκολη στην Κομισιόν. Αλλά στην πρότασή σας δεν βλέπουμε τι θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των δικαιούχων τόπου. Είπαμε τις προάλλες στο Στρασβούργο ότι άμε, μία θέση, κάθε ΜΜΕ στην Ευρώπη ε, δώσει μία θέση απασχόληση στην Ευρώπη, τότε θα, θα, δεν θα υπάρχει πια ανεργία. Αλλά άμα κάθε έψινο πρέπει να πληρώνει 10.000 ευρώ για να δημιουργήσει αυτή τη θέση απασχόληση. δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Πώς λοιπόν εσείς θα μπορέσετε να κάνετε απλούστευση μέχρι το τέλος. Δείξτε εσείς ε, ως ε, νέο μέλος ε, που ήρθατε πρόσφατα πώς μπορεί κανείς να είναι συντομότερο et de ne poser une question que concernant les régions ε, εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τις υπερπεριφερειακές περιοχές στον νέο κανονισμό κεφάλαιο 3. Έχουμε ένα δημοσιονομικό φάκελο για την αντιστάθμιση του υπερβολικού κόστους σε αυτές τις περιοχές. Πρόκειται το, για το κόστος που προκύπτει από την ε, πρόταση Σόλβε στην Κομισιόν. Τώρα εσείς αυτό το ποσό το κόψατε στο μισό. Κύριε Επίτροπε, με ποιο κριτήριο εσείς ε, αποφασίσατε αυτή τη μείωση που θα είναι καταστροφική για τις υπερ, περιφερειακές περιοχές. Τελευταίο μισό. Ο κύριος Γκουτμάνης, μισό λεπτό και μετά ο Επίτροπος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όλα εξαρτώνται και βασίζονται σε αριθμούς, αριθμητικά μεγέθη. Αν πάρετε το phasing in και phasing out σήμερα από κοινού και τα προσθέσετε, είναι 26,32 δις. Αν πάρετε τα κονδύλια σε σχέση με τις μεταβατικές περιόδους ε, στο μέλλον, είναι 38,95 δις. Αύξηση 12 δις, δηλαδή 47% για περιοχές σύγκλησης μείον 20% και για ανταγωνιστικές περιφέρειες μείον 4%. Ερώτηση μία και μόνη. Γιατί μια τέτοια δυσαναλογική σχέση, δυσαναλογία σε σχέση με αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Διότι όταν δημιουργείται μεταβατικές περιφέρειες, γιατί τότε υπάρχει μια τέτοια αύξηση σε 47%. Από τον Λεβαντόφσκι έρχομαι, επίτροπο για τα αρμόδια και τα δημοσιονομικά και βλέπετε ότι έχουμε προβλήματα περιστολών, περικοπών κονδυλίων, ακόμα και σε αυτό το τομέα. Ερώτημα, γιατί να είναι τόσο δυσανάλογη η στάση σε σχέση με τρεις διαφορετικές κατηγορίες περιφερειών. Γιατί τέτοια δυσαναλογία. Λυπούμε. Έχουμε και τον κύριο Μπλάσακ. Ε, μισό λεπτό κι εσείς παρακαλώ για να ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αιρεσιμότητα εισάγεται για να καταστήσει πιο αποτελεσματική την διαχείριση. Η πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική σε περίοδο κρίσης. Γιατί όμως έχουμε εμείς την αιρεσιμότητα και στις χώρες οι οποίες δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα και <coughs> καλύπτουν όλες τις αρχές ε, της ε, συνοχής. Μετά δεν θα έχουμε εμείς επικάλυψη ε, αν χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την γραπτή ανακοίνωση. Αυτό θα μπερδέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Έχουμε χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Όχι. Σας δίνω επίσης τρία λεπτά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Όλοι συμφωνήσαμε νομίζω για κοινού στόχου για αυτή τη στρατηγική που θέλουμε να πετύχουμε. Και όταν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να αυξήσουμε την απασχόληση, το τμήμα, το μέρος εκείνο των ε, πολιτικών μας να το αυξήσουμε για αυτούς τους στόχους. Σε όλες τις περιφέρειες με, με τα ίδια μέτρα πρέπει να δράσουμε. Είτε είναι πυκνοκατοικημένες ή άρεοκατοικημένες, δεν παίζει ρόλο. Πρόσφατα με, άλλη, με άλλο έναυσμα, με άλλη αφορμή, είχαμε κάποιε περιφέρειες τη Γαλλία που εξετάσαμε. Υπάρχουν συγκρίσιμα άρεο κατοικημένε, αλλά και πολύ πύκνο κατοικημένε περιφέρειες και έχουμε πολύ ψηλό, δυσανάλογο υψηλό ποσοστό ανεργία σε αυτέ όλε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα αίτια με υποθέτω διαφορετικά μέτρα. Ο στόχο όμω είναι κοινό στόχο για όλου και για όλα τα μέτρα. Αυτή είναι η κοινή πρόκληση. Η κοινή στοχοθέτηση τη στρατηγική τη Ευρώπη 2020 όπου με σαφέστατους στόχους πρέπει να δράσουμε που φυσικά είναι κομμένοι και ραμμένοι για στις λύσεις που υιοθετούμε σε σχέση με ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Συμφωνούμε όμω όλοι, τουλάχιστον αυτό ελπίζω, ότι συμφωνούμε ότι η δημιουργία επιχειρήσεων, νέων επιχειρήσεων, στο τελος τέλο θα συνεισφέρει να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Και εντωμεταξύ και εδώ με και πολλούς μήνες ασχολούμαι με αυτά τα παραδείγματα και ακούω ότι όλο και περισσότερο εκμεταλλεύονται αυτά τα προγράμματα οι πολίτες. Έχουμε 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και έχουμε και τυχαία 23 εκατομμύρια ανέργους. Αν σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλαμβανόταν ένας άνεργος θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα άμεσα, το πρόβλημα της ανεργίας. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό. Μπορεί να συμβεί. Δεν είναι όμως ρεαλιστικό οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης να πούμε ότι αυτό το πρόβλημα θα το λύσουν εκείνες. Γιατί τότε θα πρέπει 46.000 να προσλάβουν κάθε μια από αυτές. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουμε, να συνεισφέρουν με θετικό τρόπο. Κατά τα άλλα αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει όταν δημιουργείται ελπίδα από εμάς ως πολιτικούς προς τους πολίτες. Τους δίνουμε ελπίδες και δεν τους πούμε ότι ξέρετε θα καταρρεύσει το σύμπαν αύριο και θα καταστραφούμε όλοι. Για τις επενδύσεις όταν κάποιοι χρεώνονται και κάνουν χρέη για να υπάρξει δυνατότητα δράσης σε επιχειρήσεις δεν μπορεί να τους πει κανεί στους πολίτες αυτούς ότι αύριο θα καταρρεύσει το σύμπαν και θα καταστραφούμε δεν πρέπει να λέμε ψέματα βέβαια ως πολιτικοί αλλά να μην μεριμνούμε και λέμε συνέχεια ότι όλα πάνε στραβά και δεν μπορούν να πάνε καλά πρέπει να δείξουμε θετικές προοπτικές στους πολίτες είναι σημαντικό εδώ τουλάχιστον να ακολουθήσουμε την φιλοσοφία να βλέπουμε το ποτήρι το οποίο είναι κατά το ίμιση γεμάτο ως μισογεμάτο και να μην λέμε ότι είναι μισοάδιο. Εντάξει, με πιο αισιόδοξο τρόπο να τα περιγράφουμε. Λοιπόν, σίγουρα περισσότερο ε, μεγαλύτερες προσπάθειες και μάχη δίνεται εδώ. Αλλά αυτό είναι ο στόχο ε, που έχουμε αφοσιωθεί να επιτύχουμε. Καθημερινά πρέπει να καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έλεγα πάντα. Η δική μου κοσμοθεωρία ως, επιτρόπο, ως, επίτροπο, ως επίτροπος που είμαι δεν είναι να λέω στο τέλος της δουλειάς ότι εξοικονομήσαμε κάποια κονδύλια, αλλά όχι να λέω ότι χρησιμοποιήσαμε τα κονδύλια με αηφόρο τρόπο, ώστε στο μέλλον να είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι ο στόχος μας. Έτσι κατανοώ το έργο μου και αυτή είναι η δική μου κοσμοαντίληψη και με, ε, μια και πιέζει ο χρόνος όλες τις συζητήσεις με τους συναδέλφους και τις συζητήσεις και επαφές με τους συνεργάτες μου μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να τις εξαγάγουμε τώρα Όσον αφορά την πρώτη χώρα για την Ουγγαρία που θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, δεν θα παγώσουν οι πληρωμές, αλλά αν κάτι εφαρμοστεί, αν κάτι υλοποιηθεί, τότε από το 2013 οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις, αυτές είναι που δεν θα υλοποιηθούν. Δεν θα παγώσουν πληρωμές. Όσα, όσα έχουν προγραμματιστεί θα δοθούν. Αλλά αυτό το μέσο το εργαλείο αυτό, το οποίο το έχουμε εδώ και 20 χρόνια στους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε, είναι ένα πολιτικό μέσο, πολιτικό εργαλείο και ελπίζω ότι όταν χρειάζεται μπορεί να εφαρμόζεται. Δεν θα χρησιμοποιείται όμως ώστε να παγώνουν πληρωμές ή να διακόπτονται προγράμματα και σχέδια. Μελλοντικά, μελλοντικά κάποια πράγματα μετατίθενται, αναβάλλονται. Αλλά από σήμερα μέχρι το 2013 έχουμε χρόνια, δύο, ένα χρόνο ε, καιρό για να προσαρμόσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ε, πράγματα. Παρακαλώ αυτή τη συζήτηση όταν θα συζητήσουμε τα θέματα για τη χορήγηση απαλλαγής του 2010 να τα ξαναδούμε διότι αφενός πρέπει να ελέγχουμε και πρέπει να ελέγχουμε, από την άλλη πλευρά όμως ο θεμητός και δίκαιος στόχος είναι οι πελάτες, οι χρήστες των διαθωτικών ταμείων να μην επιφορτίζονται, να μην επιβαρύνονται με γραφειοκρατική επιβάρηση. Αυτό δεν σημαίνει εν λευκό επιταγή να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς ελέγχους. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία των πραγμάτων. Βοηθήστε με εμένα ω Επίτροπο, εσεί ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και Ανάπτυξη, να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ επιβαρύνσεων και αναγκαίων ε, ελέγχων που στο μέλλον πρέπει να υφίστανται και πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι. Για τι ελάχιστε τώρα ε, ενισχύσεις ε, ε, όταν κάνουμε λόγο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακές επιδόσεις τουλάχιστον και πρέπει να το πούμε δημιουργείται η εντύπωση ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε μορφή ελαστικότητα. Δηλαδή να λέμε 20% θα διαθέτει και όχι παραπάνω ούτε παρακάτω. 25% για το EFSF e όχι παραπάνω, όχι λιγότερα. Και Αναφέρεται όμως ελάχιστον, εδώ έχουμε την ε, ελαστικότητα, ελάχιστον τόσο της εκατό. Αν θα διατεθεί περισσότερο, ε, αυτό είναι η ελαστικότητα που θα έχουν οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Στο τέλος τέλος να αποφασίσουν αν θα διαθέσουν το ελάχιστο ή παραπάνω. Νομίζω εδώ υπάρχει αρκετό πολύ περιθώριο να δράσουμε σωστά. Και για τις μεταβατικές περιφέρειες, ενδιάμεσες περιφέρειες που ανέφερε ε, ευρωβουλευτές, οι αλλαγές αυτές απορρέουν, δημιουργούνται, μια και ο αριθμός των περιφερειών αλλάζει ως αριθμός σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Από τις 271 περιφέρειες έχουμε 84, αν θυμάμαι καλά, που είναι περιφέρειες σύγκλησης και στην επόμενη περίοδο αναμένουμε 64 64 έως 68 σε αυτή την κατηγορία. 31 δηλαδή έως 35 εκατομμύρια πολίτες λιγότεροι θα κατοικούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Και γι' αυτό η κατανομή, ο επιμερισμός για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ε, θα είναι χαμηλότερο ποσό διότι ανακεφαλήν θα πληρώνονται οι κάτοικοι αυτών των περιφερειών, θα λαμβάνουν ένα ποσό και επειδή υπάρχει αυτή η σημαντική μείωση πληθυσμού σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό διατίθεται με μικρότερο ποσό στις μεταβατικές περιφέρειες. Οι περισσότερο ανεπτυγμένε περιφέρειες σε απόλυτα μεγέθη θα παραμείνουν στα ίδια ποσά όμως η αντιστάθμιση βρίσκεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των μεταβατικών περιφερειών. Εκεί έχουμε το συν πλήν της διαφοράς. Και αυτό υπεξηγεί και την ερώτηση του συναδέλφου από τη Φινλανδία. Ο αριθμός των κατοίκων δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά το επίπεδο ΑΕΠ που έχει η επιμέρους περιφέρεια, είτε ανήκει στη μία είτε στην άλλη κατηγορία. Δεν απάντησα όλες τις παρεμβάσεις σας, αλλά ο κύριος Νίκλας Μάρτιν, θα μπορέσει να το κάνει αυτό και να συνεχίσει εξ ονόματό μου. ολοκληρώνοντα, θέλω να δραθώ την, ε, ευκαιρία να ευχαριστήσω κάποιον που για πολλά χρόνια επιτυχώς εργάστηκε για την περιφερειακή πολιτική αυτή τη στιγμή ε, αλλάζει τον πρώην ε, γενικό μας διευθυντή Γκάνερ που πραγματικά μπορώ να πω ότι βοήθησε σημαντικά τον επίτροπό του. Μέχρι την τελευταία μέρα δούλευε με αποτελεσματικό τρόπο. Ποτέ δεν εγόγγιξε, ποτέ δεν παραπονήθηκε. Σε αυτόν τον κύκλο θέλω να αποτίσω φορό τιμής ε, προσωπικά και προφορικά να ευχαριστήσω για το έργο που επετέλεσε και θα το ακούσατε ήδη. Από την 1η Φεβρουαρίου θα έχουμε ένα νέο γενικό ε, διευθυντή, τον κύριο Βάλτερ Ντεφάκου. είναι πολύ πεπειραμένο και που επί χρόνια δούλευε στην περιφερική πολιτική. Ήταν ε, μέλος ε, των διαφορετικών επιτρόπων του γραφείου διαφορετικών επιτρόπων στο παρελθόν κατά την δεκαετία του 80 ήδη. Έχουμε τι καλύτερε προποθέσει με αυτόν για να καλύψει τι ανάγκε του αξιωματικού αξιώματό του με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει κατά το επόμενο έτο διαπραγματεύσεων και εφαρμογή κανονισμών. Ευχαριστώ. Uh, you, much. And, um... Ευχαριστώ πολύ. So we will and, and we, we... Θα συνεχίσουμε και σας ε, ευχόμεθα ότι ο, ο βοηθός ε, γενικός διευθυντής σας ε, δεν θα πει ότι σφάλατε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση τώρα. Κύριοι um, Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές ο Επίτροπος αναφέρθηκε στον Νίκαλας ε, Μάρτιν που ότι θα έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τις απαντήσεις. Θα αρχίσουμε με αυτό και μετά θα περάσουμε στη συζήτηση για τα τέσσερα θέματα που αποφασίσαμε να έχουμε για τη σημερινή συζήτηση και θα εξηγήσουμε τα τι θα γίνει με τα δέκα άτομα που δεν μπόρεσαν να θέσουν ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, ένα φάσμα διαφόρων ερωτήσεων που καλύφθηκαν εν μέρη, δεν είχε χρόνο να επανέλθει σε μερικές και θα απαντήσω σε αυτές. Θα αρχίσω με το θέμα της απλούστευσης. Παρόλο που ο Επίτροπος Χαν μίλησε για την απλούστευση, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο που αναφέρθηκε ε, διότι λέχθηκε ότι δεν ασχολήθηκε ε, με τέτοια αποτελέσματα η Κομισιό ε, και κυρίως για την απλούστευση υπέρ των δικαιούχων. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Έχουμε, ε, είχαμε μια χρήσιμη συζήτηση γι' αυτό και πρέπει να μπούμε στις λεπτομέρειες, διότι μπαίνοντας στις λεπτομέρειες μπορείτε να το δείτε. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα όπου θα δείτε ότι εσταστήκαμε στις ε, προτάσεις ε, του πακέτου απλούστευσης για τους δικαιούχους. Έχουμε απλουστευμένο κόστος και επιλεξιμότητα. Έχουμε επεκτείνει την δυνατότητα ε, χρησιμοποίησης απλουστευμένης μεθόδου με απλουστευμένο κόστος και όπου υπάρχουν ωφέλη για τους δικαιούχους. Για τους κανόνες επιλεξιμότητας έχουμε ένα κοινό σώμα ε, τέτοιων κανόνων, μεγάλη αναρμόνιση των κανόνων επιλεξιμότητας που ωφελεί πολύ τους δικαιούχους. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι στον εσωτερικό έλεγχο, ε, διότι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι το άχθος ε, του εσωτερικού ελέγχου είναι προβληματικό κυρίως για τους μικρούς δικαιούχους. Έχουμε λοιπόν μια αναλογικότητα για τις, ε, τα μικρά έργα όπου δεν πρέπει να υπάρξει έλεγχος για κάθε χρόνο. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα απλούστευσης. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η Κομισιό ε, θα εκδώσει μια ανακοίνωση σύντομα που καλύπτει όλους τους ε, τομείς ε, πολιτικής του MFF, του πλαισίου αυτού, για να δείξουμε ποια, σε ποια θέματα έχουμε έχουμε δώσει τις κατάλληλες λύσεις για την απλούστευση κάτι για το CSF το οποίο αναφέρθηκε αρκετά συχνά. Όπως είπε ο Επίτροπος Χάν, τις επόμενες εβδομάδες θα συντάξουμε ένα άτυπο έγγραφο ε, που θα παρέχει τα βασικά στοιχεία που είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικά στο CSF. Όντως αυτό έχει ως βασικό στόχο τα θυλώ, δηλαδή έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε ε, καλύτερη ένταξη της χρήσης ε, των κονδυλίων. Θα μπορούσαμε να παρέχουμε γενικές κατευθυντήριες γραμμές όταν ε, τα κράτη-μέλη θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, τα ταμεία, να δουν τι μπορούν να κάνουν με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο το Κοινωνικό, ε, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Θα είναι ένα πρακτικό έγγραφο που θα είναι χρήσιμο από την άποψη αυτή. Θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία για να έχουμε ένα feedback για να δούμε αν έχουμε φτάσει στο σωστό αποτέλεσμα. Σχετικά με τους δείκτες, βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί για τον τρόπο με τον οποίο θα νομοθετηθούν καλύτερα με, σε μια πράξη κάτι εξουσιοδότηση, νομίζω. Προσπαθήσαμε να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν και ένα από τα βασικά διδάγματα είναι ότι οι δείκτες έχουν μια χρήση, συγκεντρώνομα διοποιούν τις πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά, προς πού πηγαίνουν τα χρήματα, τι έχει επιτευχθεί, ποια είναι τα αποτελέσματα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε κοινούς δείκτες, διότι μόνο αν έχουμε ένα σύνολο κοινών δικτών μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτές ε, τις ε, πληροφορίες. Είδα ε, αυτό δεν είναι εφικτό. Χρειάζεται λοιπόν κανείς ένα σύνολο κοινών δικτών για να υπάρξει αυτή η ομαδοποίηση και που συμπληρώνεται με μερικούς ειδικού δείκτες και όπως είπε ο Επίτροπος, οι κοινοί δείκτες μας δίνουν τι έχει επιτευχθεί και όχι τα τελικά αποτελέσματα που πρέπει να προσδιοριστούν ειδικά με εξειδικευμένο τρόπο. Με τους κοινού δείκτες μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για το πώς ξοδεύονται τα χρήματα και προς τα που διοχετεύονται. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Έχουμε εδώ μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την θεματική συγκέντρωση, διότι εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό, έχει διαφορετική φύση, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η ποσότητα κονδυλίων που υπάρχει για τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι για τα γενικά, για τα σημαντικά προγράμματα. Η αρχή παραμένει βεβαίως ότι η χρηματοδότηση πρέπει να είναι εστιασμένη, δεν πρέπει να είναι διάσπαρτη, διότι πρέπει να έχουμε αντίκτυπο και αποτελέσματα από τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Γι' αυτό έχουμε έναν μηχανισμό συγκέντρωσης που συνδέεται με τον αριθμό των θεματικών στόχων, που είναι αρκετά ευρύς μέσα στις έχετε προτεραιότητες επενδυτικές μέσα στους στόχους αυτούς και το πρόσθετο στοιχείο της ευελιξίας είναι ένα σύνολο προτεραιοτήτων κυρίως για το κοινωνικό ταμείο διευρύνει το πεδίο χρήσης των κονδυλίων ε, για τα προγράμματα εδαφικής ε, συνεργασίας ε, και συνδέει με τις μακροοικονομικές στρατηγικές και τα προγράμματα διαμεθοριακής συνεργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμάσουν τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Ένα τελευταίο σημείο νομίζω ότι ο Επίτροπος δεν είχε χρόνο να επανέλθει στην χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένας περιορισμός που είναι ενδογενής στην πρόταση της Κομισιόν. Δεν είναι συνολική απαγόρευση, είναι αποκλεισμό άμεσης υποστήριξης για παραγωγικές επενδύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό βασίζεται σε αξιολογήσεις, ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι καλύτερο να υποστηρίζουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ο Επίτροπος το τόνισε αυτό ε, για να δείξει πώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, και πού. Εκεί βλέπουμε έναν συλλογισμό ο οποίος μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι άμεση υποστήριξη για παραγωγικές επενδύσεις. Υπάρχει δυνατότητα για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά αυτό συνδέεται με την ε, έρευνα και την ε, καινοτομία. Δεν πρόκειται για άμεση βοήθεια για παραγωγικές επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα βασικά σημεία. Αν έχω ξεχάσει κανένα σημείο, σας παρακαλώ να μου το υπενθυμίσετε. Χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση. Κύριε Μπάσερ, με συγχωρείτε. Ε, ξέρω ότι είναι κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η διασύνδεση αυτή δεν είναι μέρος ε, του πακέτου ε, συνοχής. Είναι μια ξεχωριστή νομοθετική πρόταση της Κομισιό και η διασύνδεση είναι σε σχέση με τα 10 δισεκατομμύρια που προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής. Το σημαντικό που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτό το τμήμα του Connecting Europe πρέπει να συσχετιστεί με την χρηματοδότηση για την επίτευξη κοινών στόχων, κυρίως με τα δέκα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πρόκειται για ένα συνδυασμό ε, ε, συστημάτων ούτω ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες για την δημιουργία όλων των διασυνδέσεων που επιθυμούμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό που θεωρούμε σημαντικό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στους μηχανισμούς που εισάγουμε είναι να βεβαιωνόμαστε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προγραμματίσουν καταλήλως και σαφώς ούτως ώστε να βλέπουμε για τα βασικά προγράμματα υποδομών τι θα χρωματιδοθεί από το μέσο Connecting Europe και θα έπρεπε να προγραμματιστεί στην χρηματοδότηση με το Ταμείο Συνοχής και με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να δούμε καλά πώς γίνεται αυτή η διασύνδεση και ποια είναι η εξέλιξη της νομοθεσίας για το μέσο Connecting Europe, ούτως ώστε λειτουργικά να επιτευχθεί αυτή η στρατηγική προγραμματισμό. Ε, φαντάζομαι ότι για τα κράτη-μέλη είναι σημαντικό τι συμβαίνει με τα χρήματα που δεν επενδύονται. Αγαπητοί συνάδελφοι, οκτώ από εσά δεν κατόρθωσαν να θέσουν ερωτήσεις ε, στον Επίτροπο, ε, διότι όλοι μακρηγόρησαν. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να θέσει μια σύντομη ερώτηση από αυτόν τον κατάλογο, επειδή κρίνει ότι είναι σημαντική για τον Γενικό Διευθυντή, μπορεί να θέσει την ερώτηση. Δαλλιώς ε, θα περάσουμε στην συζήτηση που προβλέπετε. Και μετά θα μπορούμε να δώσουμε μια υπόσχεση ότι αυτός ο κατάλογος θα έχει προτεραιότητα στη μελλοντική συνάντηση με τον Επίτροπο. Περνάμε τώρα, Αραμύρα πολύ σύντομα. Είναι κρίμα, κρίμα που δεν μπόρεσα να μιλήσω κατευθείαν με τον Επίτροπο. Δέκα χρόνια ως ε, κοινοβουλευτική βοηθός ε, συμμετείχα στην ίδια συζήτηση και τα θέματα, ε, βλέπω ότι θέματα που συζητούσαμε τότε δεν έχουν ξεπεραστεί. Οι δείκτες, η συνοχή, το θέμα της συγκέντρωσης ή όχι των κονδυλίων. Στην προκειμένη περίπτωση η Κομισιόν θα έπρεπε να απαιτήσει μία πραγματική αξιολόγηση των διαφόρων συμφωνιών, συμβολέων κλπ. με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν περιφερειακές οντότητες με νομοθετική υπόσταση. Το είπε αυτό και ο Επίτροπος. Θα έπρεπε λοιπόν να επιμένουμε επειδή η συμμετοχή αυτών των περιφερειών δεν ήταν εγγυημένη στο παρελθόν, να επιμένουμε ούτως ώστε να επιτευχθεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι η εμπλοκή τοπικών ε, τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών σε όλη αυτή την ιστορία θα βοηθήσει και στη σωστή διαχείριση των κονδυλίων. Πάντοτε είχαμε τέτοιους μεγάλους ε, και ευρύς ορίζοντες που δεν φτάνανε ποτέ σε τοπικό επίπεδο ε, μεγάλα σχέδια αεροδρομίων ή σχέδια καθαρισμού του νερού κτλ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω ότι έχετε μια ερώτηση, έτσι δεν είναι, λέει πρόεδρος. Εγώ έρχομαι από τη Γαλλική. Θεωρούμε ότι οι δείκτες που έχουν οριστεί δεν είναι πάντα οι καλύτεροι για να μπορέσουν να εγγυθούν την σύγκληση. Θέλω να ξέρω λοιπόν ποια είναι η, κομισιο, η θέση της Κομισιόν για τις μεταβατικές ε, περιφέρειες. Και επίσης τι γίνεται με το κριτήριο της καταπολέμησης της ανεργίας. Ξέρουμε πόσο υποφέρει από αυτήν τη μάστιγα. Καταλαβαίνω. Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε, οι κατηγορίες ε, των ε, περιφερειών. Αν θέλετε σύντομα να απαντήσετε ή το κρατάμε για την συζήτηση και να απαντήσετε αργότερα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πρώτος. Έχουμε τέσσερα θέματα. Η εισαγωγή σε δύο θέματα θα γίνει από τον Λαμπέρτα Μίστερολ και δύο θέματα από την ε, Κωνσταντσα ε, Κρέλ. Αρχίζουμε με την Κωνσταντσα Κρέλ. Φαίνεται. Κωνσταντσα, μπορείτε τότε να μας εισαγάγετε τα δύο θέματα που συμφωνήσατε με το Λαμπέρ για την εισαγωγή. κυρία Κρέλ, θα το προσπαθήσω. Θα ξαναξεκινήσω με το αγαπημένο θέμα της ελαστικότητας και των ποσοστώσεων. Λοιπόν, λοιπόν εξεπώνησα ένα πίνακα επισκόπησης, ανασκόπησης. Πώς η ελαστικότητα επιτρέπεται και βρίσκεται στις επιμέρους περιφέρειες με αυτή την κατηγοριοποίηση. Και αν κινούσαμε από αυτό το στοιχείο, ο κύριος Επίτροπος Χάν είπε ότι είναι ελάχιστα ποσοστά όλα αυτά. Δηλαδή μπορούν να δαπανηθούν μεγαλύτερα κονδύλια, περισσότερα κονδύλια για αυτούς τους στόχους. Όμως εδώ έχουμε το θέμα της ελαστικότητας και για τους στόχους που δεν καλύπτονται. Τι γίνεται οι εταίροι στις συζητήσεις με τους οποίους εγώ έχω συζητήσει και συζητώ και που προέρχονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί όλοι να κάνουν λάθος και να μου έχουν δώσει όλοι λανθασμένα στοιχεία. Τι να πω, και να μην έχουν πετύχει την ουσία του θέματος. Όλοι όμως μου λένε ότι η θεματολογική επικέντρωση εντάξει είναι κάτι σωστό. Δεν πρέπει όμως αυτοί οι στόχοι να περιγράφονται με αυτόν τον τρόπο όπως έχουν συμπεριληφθεί. Βλέποντας τώρα τις ε, περιφέρειες σύγκλησης και που υπάρχει σχετικά περιθώριο για την προσαρμογή. Το θέμα της ε, συμπίκνωσης θεματολογικά δεν είναι τόσο έντονο, αλλά το συνολικό ποσό από τις προτάσεις που έχουν γίνει για τους πόρους είναι 40% ακόμα ελεύθερα διαθέσιμο για τις ιδιαίτερες προτεραιότητες ε, των περιφερειών και των κρατών μελών. Στις μεταβατικές όμως περιφέρειες, στη μεταβατική κατηγορία περιφερειών, μόνο 20% είναι αυτό το ποσοστό το οποίο μπορεί έτσι να διατεθεί. Στις πιο ανεπτυγμένες, καλύτερα ανεπτυγμένες περιφέρειες ως κατηγορία είναι μόνο περίπου 17-18% αυτό το ποσοστό. Τι βλέπουμε. Όλα αυτά δεν επαρκούν, πιστεύω εγώ. Δεν επαρκούν αυτά τα ποσοστά. <clears throat> δεν καλύπτεται το θέμα ή δεν αναφέρεται καν ή πολύ στο περιθώριο καλύπτεται όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα δημογραφικές λέει εξελίξεις να τις αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο. Πού αντανακλάται αυτό κάπου. Πουθενά δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες αυτό. Διότι υποτίθεται ότι όλες οι προτεραιότητες ω στόχοι πρέπει να συνεισφέρουν να αντιμετωπιστεί η δημογραφική αυτή φθήνουσα εξέλιξη, η υπεργύρανση. Αλλά δεν επαρκούν αυτά τα οποία προτείνονται με κανένα τρόπο. Και όταν λέμε αφενός Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Από την άλλη πλευρά δεν αφήνουμε περιθώριο για να δράσουμε ή αντιδράσουμε σωστά τι μπορεί να γίνει διαφορετικά στις περιφέρειες. Σε μια περιφέρεια, για παράδειγμα, της Ισπανίας ή άλλης χώρας είναι πολύ διαφορετική από ό,τι σε μια γερμανική περιφέρεια ή πολωνική περιφέρεια. Παρότι το ίδιο πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε όλες αυτές τις περιφέρειες αλλά με διαφορετική ένταση σε διαπραγμάτευση λοιπόν με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες πρέπει να καταλήξουμε σε περισσότερη ελαστικότητα, μεγαλύτερη ευελιξία εδώ. Θα το πετυχαίναμε αυτό για παράδειγμα αν λέγαμε με το ESF <clears throat> e έχουμε μια πολύ μεγάλη επικέντρωση, συμπίκνωση κονδυλίων σε συγκεκριμένες στοχοθετήσεις. Όταν λέμε τουλάχιστον 25% ESF, ε, τότε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό να κοιτάξει κανείς όμως στη συνέχεια αν μια περιφέρεια μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση της φτώχειας που αντιμετωπίζει να βελτιωθούν οι συνθήκες ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να γίνουν προσφορές και μέτρα για την κατάτηση και εκπαίδευση εργαζομένων. Αλλά αυτά οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τις περιφέρειες. Είμαι πεισμένη ότι οι περιφέρειες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για όλα αυτά. Γι' αυτό οι απαιτήσει από πλευρά μια περιφέρεια μπορεί να είναι ναι, χρειαζόμαστε 50% ESF. Σε άλλε περιφέρειε μπορεί να χρειάζονται 30% μόνο ESF και ίσως στο τέλος τέλος έτσι μπορεί να απορρεύσει να δημιουργηθεί μια εικόνα. Μια εικόνα που πιθανότατα δεν θα είναι και τόσο δραματικά διαφορετική. Αλλά όμως το θέμα της θεματολογικής ε, επικέντρωσης που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να είναι ένας στόχος, αλλά πρέπει να υπάρχει και περιθώριο διαπραγματεύσεων για τις περιφέρειες σε ένα πιο ευέλικτο, πιο, πιο ελαστικό πλαίσιο. Και θα ήθελα, αν γίνεται, απλά να συζητήσουμε Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να γίνει αυτό. Και αισθάνομαι, πώς να το πω, όπως αν ήμουν μαθήτρια σε μια τάξη στο σχολείο και μου έλεγαν «Α, αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσει. Μπορεί όμως να δοθούν και περισσότερα για αυτό το στόχο. Ε, στο τέλος τέλος τι γίνεται. Φτάνουμε στο 100% και δεν μπορούμε να διαθέσουμε παραπάνω. Και όταν λέμε ότι αντί 300 ε, τόσα δισεκατομμύρια θα διατεθούν 500 δισεκατομμύρια, ε, τότε εντάξει να συζητούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη επικέντρωση θεματολογικά, διότι τα περιθώρια θα ήταν πολύ μεγαλύτερα λόγω της αύξησης των ποσών. Αλλά αυτό δεν γίνεται εδώ. Τέτοιου είδους ελαστικότητα δεν θα, δια... θα είναι διαθέσιμη, φοβούμε. Το αντίθετο φοβούμε ότι θα γίνει. Θα είναι πιο πιεστικά τα περιθώρια λόγω περιορισμένων κονδυλίων. Πρέπει να δούμε εδώ πώς μπορούν τα συμφέροντα των ίδιων των περιφερειών και των κρατών μελών που εμείς ως Ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε μπορούν να ληφθούν υπόψη και των κατανοητών συμφερόντων που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξευρεθεί ένα συμβιβασμός. Μία οδός συμβιβαστική όπου και τα δύο μπορούν να συνδυαστούν και να γίνει ένα διάλειμμα, να υπάρξει μία ανάσα που θα πάρουμε για τη σωστή πολιτική συνοχής που θα ακολουθήσει τη σωστή πορεία ώστε να μπορούν στοχοθετημένα να υποστηρίζονται οι περιφέρειες προς το συμφέρον συμφέρον της στρατηγικής του 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς το συμφέρον τους. Αυτά για την ελαστικότητα και για τις ποσοστώσεις, για το θέμα της απλούστευσης. Ίσως θα έπρεπε το θέμα σήμερα σχετικά σύντομα να το συζητήσουμε διότι γνωρίζω ότι στις 20 Μαρτίου θα έχουμε μία ακρόαση που θα διεξαχθεί για αυτό το θέμα έντονα και σε βάθος ασχολήθηκα και εξέτασα τις προθε... προτάσεις που στον γενικό κανονισμό εμπεριέχονται και έκανα μια πρώτη προσέγγιση να δω πώς ε, για τον κανονισμό, για το ειδικό ταμείο προβλέπονται αυτές οι προτάσεις. Έχω την εντύπωση όταν σε βάθος πολύ ε, σε λεπτομέρειες εξετάζει κανείς αυτά και κατανοεί τι γίνεται σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό από διάφορες πλευρές, τότε ουσιαστικά η Επιτροπή έχει κάποιες πολύ ευφυείς προτάσεις που κάνει και στη διαχείριση και στην λειτουργία που προβλέπεται να απλουστευτούν κάποια πράγματα με αποτελεσματικό τρόπο. Καλό θα ήταν, θα έλεγα, αυτές τις επισημάνσεις, για παράδειγμα την ετήσια έκθεσης προόδου, που σε τρία διαφορετικά σημεία αναφέρεται αυτό. Το ότι δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι η βάση, τα θεμέλια. Να πούμε εντάξει ακούστε το άρθρο τάδε, δεν ξέρω αν αληθεύει, το 45 ας πούμε το άρθρο 45 στο Γενικό Κανονισμό. Λέει αυτό και αυτό αυτό και το άλλο. Και όταν πάμε στον εξειδικευμένο κανονισμό να αναφερόμαστε σε αυτό το άρθρο στο 45. Να μην νομίζει κανείς ότι πρόκειται για άλλη ξεχωριστή έκθεση πρόοδου. Να ξέρει ότι πρόκειται για το ίδιο άρθρο. Γιατί διαβάζοντας κανείς τα πράγματα έχει κανείς την εντύπωση ότι ο αριθμός των εκθέσεων που θα υποβάλλονται θα είναι υπερβολικά αυξημένο στο μέλλον ο αριθμός των εκθέσεων. Και αν το διαβάζει κανείς προσεκτικά βλέπει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δίνει λοιπόν τη δυνατότητα μείωσης εκθέσεων απλούστευσης του αριθμού, αμείωσης του αριθμού των εκθέσεων. Υπάρχει ένας κίνδυνος θα έλεγα να υπάρξουν κάποια σημεία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγε να τα διαμορφώσουμε με πιο απλό τρόπο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συμπράξουν εδώ. Και υπάρχει, πιστεύω, φοβούμε ο κίνδυνος, υφίσταται ο κίνδυνος στα κράτη-μέλη να αφαιθεί ένα περιθώριο τη δική τους γραφειοκρατία να την επεκτείνουν, να την επεκτείνουν περαιτέρω, λέγοντας «Α, εδώ ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθούμε εδώ, εμείς οι ίδιοι, τα κράτη-μέλη». Να λοιπόν γραφειοκρατία. Να καθοριστεί λοιπόν σε ένα εδάφιο, σε ένα τμήμα ή σε ένα παράρτημα ή σε μια delegated act, σε μια κατεντολή πράξη, έναν ορισμό, ένα προσδιορισμό του τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε. Και σε αυτό το πλαίσιο θα με ενδιέφερε πραγματικά έντονα να μάθω τι είναι αυτό ουσιαστικά, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κανονικής ετήσιας έκθεσης προόδου και εκείνων των εκθέσεων προόδου που αφορούν το 2017 και 2019 και θα συνταχθούν τότε, ιστερότερα; Ποιες ποιοτικέ διαφορές υπάρχουν στις πληροφορίες που θα εμπεριέχονται στις επόμενες εκθέσεις σε σχέση με τις προηγούμενες. Δεν βλέπω ποια θα ήταν αυτή η διαφορά. Δεν το κατανοώ από τους ορισμούς αλλά έχω την αίσθηση ότι εύκολα θα μπορούσε να καταλήξει κανείς την πεποίθηση ότι όταν γίνονται κάποιες εκθέσεις αξιολόγησης, ε, παίρνουμε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης και εννοούμε ίσως ότι δεν θα χρειαζόντουσαν αυτές οι, εκθέσει οι εκθέσεις προόδου 2017-2019. Υπάρχουν περιθώρια λοιπόν για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό που θα είναι σημαντικό είναι το θέμα της απλούστευσης. Σε αυτό το θέμα οι προτάσεις που στον γενικό κανονισμό διατυπώνονται και στους επιμέρους κανονισμούς των ταμείων να εφαρμόζονται και να ε, ε, συμμορφωνόμαστε με αυτούς. Μετά από πρώτες συζητήσεις για το γεωργικό τομέα, τον τομέα της κοινή αγροτικής δημοτικής πολιτικής όπου σε αυτόν τον γεωργικό τομέα νέες απόλυτα καινούριε απαιτήσει για νέε εκθέσει διατυπώνονται που ίσως δεν χρειάζονται στον αγροτικό τομέα και ίσως μάλιστα επιδεινώνουν τα πράγματα σε σχέση με τις, τον αριθμό εκθέσεων που συντάσσονται. Από την άλλη όμως πλευρά, στον τομέα της διαφορετικής πολιτικής υπάρχουν κάποια καινούργια πράγματα, τα οποία σημαίνουν και συνεπάγονται μικρότερη επιβάρηση, λιγότερα βάρη. Πρέπει να μην υπάρχουν μεταθέσεις μεταξύ των ταμείων και παρεκκλήσεις που θα δημιουργούν δυσχέρειες παρότι μια κοινή διοίκηση και διαχείριση θα διευκόλυνε τα πράγματα διοικητικά ή διαχειριστικά. Μια τελευταία παρατήρηση. Μου βλέπω να λείπει η αποφασιστική ένδειξη ότι εκείνοι που πραγματικά συντάσσουν τις, ε, τα αιτήματα και είναι οι εποφελούμενοι στο τέλος τέλος θα πρέπει να συντάσσουν αιτήσει επί αιτήσεων. Νομίζω πρέπει να υπάρχουν απλουστεύσεις στο σύστημα διαχείρισης, στο σύστημα ελέγχων. Δεν βλέπω όμως πραγματικά να υπάρχουν απλουστεύσεις για εκείνους που θα υποφελούνται και θα πρέπει να συντάσσουν αιτήσει και που θα υποβάλουν αιτήσει και που στη συσσόρευση ή προσθήκη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών γραφειοκρατικών συστημάτων θα αποτελούν συσσόρευση. Και στο τέλος θα πούν αυτοί οι άνθρωποι αφήστε μας ησυχού. Είναι τέτοια η γραφειοκρατική επιβάρηση που δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω. Δεν βλέπουμε να γίνεται αυτή η απλούστευση εδώ, διοικητικά και διαχειριστικά εδώ. Θα πρέπει ο Γενικός Κανονισμός πιο εξειδικευμένα να προβλέπει τέτοια διευκόλυνση και ελάφρυνση. Και η ισοπεδωτική αυτή καθολοκληρία συλλήβδη αντιμετώπιση μόνη τη δεν επαρκεί. Πρέπει πιο εξειδικευμένα να γίνουν πράγματα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτά εισαγωγικά. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ σύντομα, διότι πιστεύω ότι υπάρχει έντονος συσχετισμός μεταξύ των διαφορετικών παραγράφων και έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα αρκετές φορές, έχουμε δει το κείμενο βλέποντας το κείμενο για τις ερμηνείες και τη στοχοθέτηση και το πώς ερμηνεύουμε κάποια πράγματα. Σε σχέση με τη συζήτηση, αν θέλουν να αντιδράσουν οι συνάδελφοι σε αυτό, είναι για την κατηγορία των περιφερειών η παρέμβαση. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να ε, το εξετάσουμε δεν είναι ε, κάποια επανάληψη σε σχέση με την πέμπτη έκθεση για τη συνοχή παρότι στο τέλος της συζήτησης σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριο Χάν σήμερα, τι θα γίνει αν πέσει, καταρρεύσει το σύμπαν ή καταρρεύσει ο κόσμος, τι θα συμβεί αν, στο τρομερό αν. Ε, λοιπόν, έχουμε όλο και λιγότερα κονδύλια, δεν ακολουθούμε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν. Σωστό λοιπόν είναι να σκεφτούμε τους στόχους της Ευρώπης, ε, της στρατηγικής Ευρώπης για το 2020. Πρέπει να είναι μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για κάθε περιφέρεια και πρέπει να είναι κομμένη και ραμμένη η πολιτική μας για τις ανάγκες των περιφερειών. Και με την προσέγγιση των ποσοστών ε, του ΑΕΠ έχουμε αυτή την προσέγγιση από πλευράς μας. Αυτή είναι η θέση που έχουμε σήμερα και η αφετηρία. Δεν να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση από μηδενικό σημείο για το έβδομο σημείο. μακροοικονομική όροι και προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν όλα αυτά είναι ένα ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα θέμα. Μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε περισσότερα από όσα έχουν ενταχθεί και προβλέπονται από πλευρά του Πράσινου Ταμείου ήδη. Αλλά είναι ένα εκ των άνω, αυτό μια εκ των άνω πρωτοβουλία. Κάνοντα ε, βήματα για τα επόμενα ταμεία, τα άλλα ταμεία, περιπλέκονται περισσότερα τα πράγματα και στη Γεωργία και στο δεύτερο πυλώνα και για την ανάπτυξη τη υπαίθρου και όλα αυτά. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, πολύ πιο σύνθετα εκεί. Εμείς στο έγγραφό μας έχουμε σαφώς διατυπώσει ότι δεν θεωρούμε ότι έχουμε εδώ ε, συνάφεια, συνάρτηση των δύο ε, ε, αυτών αξώνων ή επιπέδων και αυτό ξενίζει και θα πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπε η Κωνσταντσε, οι σοσιαλιστές είναι εναντίον. Εγώ ως εισηγητής είπα θα δω ποια τελική πρόταση θα υποβληθεί. Μέχρι σήμερα δεν βλέπω όμως να υπάρχει ο, η ορθολογική σκέψη που να τα επεξηγεί όλα αυτά. Είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε με τους συναδέλφους στην ομάδα των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό είναι κάτι που έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εκείνοι που το επινόησαν και το ε, συνέταξαν αυτό πρέπει να δώσουν τα επιχειρήματα. Είναι δουλειά της Προεδρίας, είναι δουλειά του Συμβουλίου να μας εξηγήσουν πώς θα πρέπει να διαμορφώσουμε διαμορφωθεί συζήτηση το επόμενο εξάμεινο. Και οι όροι και προποθέσει εξ άντε, αυτό είναι κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, διότι δίνει εξουσία, δίνει σάρκα και οστά, περιεχόμενο στην εταιρική σχέση. Πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ γοργά ήδη κατά τα τέλη του έτους και μέσα στο 2013 πρέπει να υπάρξουν αυτές οι συμβάσει εταιρικής σχέσης στο τραπέζι έτοιμες είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει τα σχόλιά μας. Είναι σχόλια υπό τον όρο του πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Εμείς θα έχουμε μια κρόαση για όλα αυτά και θα ακούσουμε, θα εισακούσουμε τις απόψεις των μελών. Και υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τι ιδιαίτερότητε και τι συστάσει όσον αφορά τα κράτη και τι περιφέρειες. Και υπάρχει και συσχετισμό σε σχέση με τη συζήτηση που διεξήχθη για την ελαστικότητα, την ευελιξία. Προ αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να κινηθούμε επίση, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να επενδύσουν προ την ίδια κατεύθυνση, διότι εμεί κάνουμε λόγο για κονδύλια συνοχή για τη στρατηγική του 2020, όμω θα υπάρχουν πολλά περισσότερα κονδύλια τα οποία θα δίνονται από τα κράτη-μέλη, επιχειρήσει επιχειρήσεις, δραστηριότητε δράσεις, καινοτομία και όλα αυτά. Όχι μόνο συζητούμε λοιπόν αυστηρά για το πώς θα διαθέσουμε εμείς τα κονδύλια μας, αλλά αντίθετα έχουμε και αμφίδρομα εδώ δυνατότητες δράσης. Θα υπάρξουν χρήματα και από αλλού. Πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει μια σαφής προοπτική για τις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας, ώστε τα κράτη-μέλη εθνικά να μπορέσουν να δράσουν και από πλευρά τους. Δεν είναι μόνο ότι δίνουν κάτι, δίνουμε κάτι, αλλά ζητούμε και κάτι από τα κράτη-μέλη. Και η τελευταία μου παρατήρηση αφορά τις ε, εταιρικέ αυτέ σε συμβάσεις ή συμφωνίες. Ακούγοντας τις συζητήσεις σήμερα, ακόμα μου φαίνεται ότι γίνεται λόγος και στρέφουμε τέτοια προσοχή στα κράτη-μέλη και μετά α, λέμε «Α, εντάξει, Εσεί θα αποφασίσετε τι θα γίνεται με τι ε, περιφέρειε και τα αστικά κέντρα και τι πόλει, πώ θα ενταχθούν. Δεν μ' αρέσει κάτι τέτοιο όμω. Γι' αυτό θέλω να τονίσω την ιδέα να έχουμε ένα έγγραφο ξεκάθαρο που θα ξεκινεί και θα θέτει όρου και προποθέσει εξάντε, εκ προημίου. Τι κάνει κάθε χώρα, τι κάνει, πώς εμπλέκει του κοινωνικού εταίρου ένα κράτο κομμένη και ραμμένη πολιτική και προγράμματα. Τι θα γίνει ευθύ εξ αρχή να το ξέρουμε. Και όχι να λέμε θα το κάνουν αυτό, κάτι το δοκούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρχει μεγάλη πίεση χρηματοοικονομικά, αλλά κάποτε στο τέλο του 2013 θα βρεθούν όλοι υπό μεγάλη πίεση, δεν θα δρουν συντονισμένα σε ένα ενίο πλαίσιο. Δεν είναι αυτό που θέλουμε καλά προετοιμασμένο και σχεδιασμένο. Πρέπει πολλά να γίνουν λοιπόν σε σχέση με αυτά τα σημεία και σε σχέση και με το έγγραφο που πρέπει με αυτό το οποίο έχει, έχουμε σήμερα στα χέρια μας να αποσαφινιστούν πολλά σημεία για να σημειωθεί πρόοδος. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα με τους συζητητές που θέλουν να μιλήσουν ακολουθώ ότι τον κατάλογο, αλλά δεν χρειάζεται όλοι να μιλήσουν διότι εστιαζόμαστε ε, στα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε ότι και στον Γενικό Διευθυντή ότι δεν μην ρωτήσουμε την DG Regio για το νέο μέσο. Η απάντησή σας είναι πολύ διπλωματική και βεβαίως ξέρουμε τι συμβαίνει και η DG Transport μας παρουσίασε την άποψη ότι έχουν τη νέα προσφορά για τις χώρες της συνοχής. Αυτή η ρητορία που είναι για την εσωτερική συζήτηση δύσκολη της Κομισιό 40 ε, δισεκατομμύρια είναι στο πακέτο συνοχής. Αυτό είναι στη συνοχή. Εάν είναι στη συνοχή, ε, το θέμα ποιος είναι υπεύθυνος ε, κλπ είναι ένα ε, θέμα στην Κομισιό, όχι σε εσά, διότι αν μιλάμε για την θεματική συγκέντρωση, θα ήθελα να πω ότι έχουμε τρία ε, ε, σημεία θεματικής συγκέντρωσης. Πρώτα απ' όλα ESF, 25% είναι θεματική συγκέντρωση. Δεύτερον, το μέσο που είναι ε, θεματική συγκέντρωση. Τρίτον, ε, το ERDF, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και τέσσερα, μέσα στο ESF έχουμε και πάλι θεματική συγκέντρωση. Υπάρχει πάρα πολύ θεματική συγκέντρωση μέσα. Ε, σας παρακαλώ, αν τα βάλετε όλα μαζί, η ευελιξία μειώνεται όλο και περισσότερο. Αυτή ήταν η αντίδρασή μας σύμφωνα με την απλούστευση, όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, είναι, είμαστε πάρα πολύ ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το CSF αλλά και για το περιεχόμενο. Το καθεστώς είναι ένα πράγμα, αλλά το περιεχόμενο είπαμε και στον Επίτροπο ότι ε, μπήκατε τόσο πολύ στις λεπτομέρειες για τις στρατηγικές προτεραιότητες, θα είναι τώρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν δράσεις, διότι έχετε δράσεις και προτεραιότητες ή πρέπει οι προτεραιότητες να είναι πιο γενικές ή απαραίτηστε από τις δράσεις. Δεν, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα προχωρήσετε. Και αυτό είναι το ίδιο με τις συμβάσεις εταιρική σχέσης. Έχουμε το πρόβλημα του οδοντολογικού κώδικα αν θα είναι το γενικό στοιχείο ή όχι και βεβαίως ε, τα στοιχεία των ε, δικτών που συνδέονται με τη θεματική συγκέντρωση. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ένα είδος ε, δικτών. Αλλά είναι δίκτες που συνδέονται με τι. Είναι δίκτες για τα θεματικούς στόχους ή δίκτες για τις επενδυτικές προτεραιότητες ή δίκτες για τις δράσεις κλειδιά από ό,τι καταλαβαίνω, είναι οι δείκτες ε, για τα output, για τα, αποτελέσματα. Ως αποτέλεσμα είναι ότι ο κατάλογος ε, των δικτών ως νομοθετική πράξη θα δημιουργήσει πάρα πολύ σύγχυση. Πρέπει να υπάρχουν κοινοί δείκτες. Πρέπει να δείτε αν θα υπάρξει νομοθετικό κείμενο, διότι θα διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο τους δείκτες. Αυτή είναι η νομοθεσία. Ε, πρέπει να δούμε αν θα συζητήσουμε τους δείκτες ή όχι. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα λέγονται εδώ στο κείμενό μου. Και δεν ήταν το θέμα το σημερινό. Αν θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα της, ε, του περίφημου καταλόγου των πόλεων που πρέπει να είναι αστικές περιοχές και το 5% ε, δεν είναι 5% επιπλέον, είναι 5% μέσα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοείται με αυτό και βεβαίως η αστική πλατφόρμα. Διότι όταν συζητάμε στη, στη Γενική ε, Διεύθυνση, όταν έχετε τις λογικές συνέπειες, ε, τον κατάλογο των αστικών περιοχών ε, με βιώσιμη ανάπτυξη, έχετε αστική πλατφόρμα. Όλα αυτά είναι λογικά. Αλλά σε πάρα πολλέ παρουσιάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν παρουσιάζονται έτσι τα πράγματα. Έχουμε διαφορετικά μηνύματα που μας έρχονται από την Κομισιό. Ίσως δεν είναι θέμα για σήμερα, αλλά είναι σημαντικό το θέμα. Πρέπει να έχουμε ένα σαφές μήνυμα. Σήμερα πήρα ε, την ε, πληροφορία από την Επιτροπή Πληροφοριών. Είναι αντίθετη προ την αστική πλατφόρμα. Δεν ξέρω, ε, νομίζω ότι σφάλουν, αλλά Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε κατά της θεματικής συγκέντρωσης, αλλά είναι και το θέμα της ευελιξίας, διότι πάμε πολύ μακριά και αναλαμβάνουμε ε, πολύ ευθύνη, πολύ ευθύνη η Επιτροπή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη ευελιξία. Αλλά όχι οτιδήποτε, ό,τι θέλετε. Έχετε επιλογή, αναλαμβάνετε ευθύνη, διαπραγματεύεται κανείς με την Επιτροπή, έχουμε μια συμφωνία ίσως για την εταιρική σχέση. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτά είναι τα στοιχεία που ήθελα να τονίσω, υπάρχουν και πολλά άλλα. Δεν ζητώ τώρα την απάντηση αλλά όσον αφορά το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πεδίο παρέμβασης υπάρχει ευξημένο ενδιαφέρον. Δεν θέλω να συζητήσω για καπνό. Ας αφήσουμε το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει το πρόβλημα με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές για το ICT και τις βασικές υπηρεσίες. Τι εννοείται με βασικές υπηρεσίες. Ε, και λέτε ότι μπορώ να καταλάβω ε, την, την οδοπία, αλλά το ICT ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση για το θέμα αυτό μεταξύ των ειδικών. Και με αυτή την απόφαση δεν θα έχουμε τις απαντήσεις για το κλίμα. Αλλά δεν είμαι ειδικό. Ευχαριστώ. Κύριοι, πρέπει να θυμόμαστε ότι ότι το ICT εκεί η επιλεξιμότητα βασίζεται σε ορισμένα στοιχεία, στην αγορά. Η αγορά υπάρχει. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Θα ήθελα να σας ζητήσω δύο πράγματα και πάλι Φαίνεται ότι έχουμε πολύ χρόνο, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές, σας παρακαλώ να είσαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι και να εστιάζεστε στα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Αυτό είναι ένα γενικό σχέδιο. Τώρα θα προχωρήσουμε με τους εισηγητές και μετά θα περάσουμε στους κοιόδης. Ο κύριος Μπουστινάρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση των δύο συνηγητών για τους γενικούς κανόνες και το έγγραφο του κ. Όλμπριν και υποστηρίζω πλήρως τις ιδέες αυτές. Μπορώ να προσθέσω ένα στοιχείο σχετικά με την μακροοικονομική σταθερότητα. Ε, στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου που προτάθηκε ε, η ε, Δημοσιονομική Ένωση όπως λέχθηκε, με στόχους που είναι όχι μόνο δεσμευτικοί, αλλά ε, στοιχεία του συνταγματικού πλαισίου όλων των κρατών, όχι μόνο της Ευρωζώνης, πιστεύω ότι τα κριτήρια που αναφέρονται στην μακροοικονομική σταθερότητα όχι μόνο επικαλύπτονται με τα άλλα, έχουμε επίσης το six-pack που είναι τμήμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Γιατί να τιμωρείτε μόνο η πολιτική συνοχή και να αντιμετωπίζετε με τον τρόπο αυτό. Επανέρχομαι ε, στην έκθεση συνοχή. Βεβαίω ε, έχουμε το μέσο Connecting Europe, διασυνδέοντα την Ευρώπη. Και είναι μέσα στο, στην έκθεση συνοχή. Πάρα πολλά θέματα ήδη Αναφέρθηκαν από πολλούς συναδέλφους, ο κύριο Όλμπριχ περισσότερο από όλους αναφέρθηκε στα θέματα αυτά. Αλλά θα προσθέσω και άλλες απόψεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να πάρουμε 10 δισεκατομμύρια ε, ε, ευρώ με, λόγω των κριτηρίων που δεν είναι ευνόητα και δεν είναι εύκολο να γίνουν αποδεκτά. Δύο, σχετικά με το management. Πώς θα βάλετε μαζί ε, ε, συγκεντρωτική ε, διαχείριση με τμήματική. Η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική. Τρία. Σχετικά με την αρχή που προτείνεται από την Κομισιό, ο πρώτος που έρχεται εξυπηρετείται. Δεν πρόκειται εδώ για λαχείο δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την ιδέα ότι ο πρώτος που έρχεται εξυπηρετείται πρώτος, διότι αυτό μπορεί να είναι δυσμενές κυρίως για τις χώρες που έχουν τις περισσότερες ανάγκες ε, τα, τα κράτη-μέλη του Ταμείου Συνοχής. Κάτι πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε να το δεχθούμε αυτό και να ψηφιστεί στην Επιτροπή και αργότερα στην, ε, στο Κοινοβούλιο και να υπάρξει και διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και πάλι για την ε, ενεργειακή απόδοση στα νοικοκυριά. Όπως είπα προηγουμένως, ζητώ να δοθεί η δυνατότητα αυτό το ειδικό κεφάλαιο να είναι ανοιχτό και για το Ταμείο Συνοχής, διότι έχω υπόψη μου ορισμένα σημεία κλειδιά είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθηθούν έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι προφανές, είναι η τοπική ανάπτυξη που χρειάζεται την περισσότερη προσοχή μας. Ε, υπάρχει προσβασιμότητα κοινωνική για την ενέργεια όταν οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται ραγδαία κάθετα και οι δυνατότητες των μεσαίων νοικοκυριών μειώνονται μεγάλο κοινωνικό κόστος. Και αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε ότι η δυσφορία ε, στην Ρουμανία οφείλεται και σε αυτές τις τιμές. Τρίτον, είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζετε τις εκπομπές αερίου, αερίου και, να να ασχοληθείτε με τους στόχους 2020, να προβλέψετε κυρώσεις εναντίον των κρατών μελών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσει που έχουν δεχθεί προτού διαπραγματευτούν την ένταξη. Πέμπτο, είναι καλό διότι θα γίνει η ενέργειά μας πιο πράσινη, πιο φιλική προς το περιβάλλον, θα μειώσουμε το κόστος και θα βελτιώσουμε το ενεργειακό μείγμα. Το γεγονός ότι δύο επίτροποι είναι υπέρ και η δήλωση του Επιτρόπου Χάν νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετική και σήμερα το πρωί η Δανική Προεδρία επιβεβαίωσε την προθυμία να υποστηρίξει την ιδέα και θα ήμουν έτομος να ενσωματώσω στο έγγραφό μου που θα έχω για την επόμενη συνεδρίαση αυτή την πρόταση. Και τέλος, <coughs> δεν έχω ακόμα λάβει σαφή απάντηση από τον Επίτροπο ε, και βιαζόταν στο ταξίδι του στο Βουκουρέστι. Θέλουμε έναν σαφή ορισμό σχετικά με τις αιρεσιμότητες, πού και πότε το Ταμείο Συνοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις όπου η αρχή του την αποτυγχάνει. Ο Επίτροπος Πότοσνικ είναι έτοιμος και είμαι πεπισμένος όχι μόνο η Επιτροπή Περιφερειών αλλά και αυτή η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και κριτήρια οδηγίας μπορούμε να το δεχτούμε αυτό γιατί αλλιώ ανοίγουμε την πόρτα για κάτι που δεν είναι και τόσο προφανές ότι είναι μέρος της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ και για την επόμενη συνεδρίαση ε, θα σας υποβάλω το πλήρες ε, πακέτο. Άλλη μια φορά διευκρινίζω. Θα έχουμε στο μέλλον συνεδριάσεις ε, για τα, τις ατομικές εισηγήσει για τα διάφορα κανονιστικά μέσα για όλα τα ταμεία. Σήμερα συζητούμε βάσει της πρότασης που προέρχεται από τους εισηγητές για γενικούς κανονισμούς, για οριζόντια θέματα αφήνοντας δυνατότητα στους τομεακούς εισηγητές τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε αυτά τα οριζόντια θέματα που επηρεάζουν ε, ή συνδέονται με τους κανονισμούς τους και σήμερα ασχολούμεθα με την ε, συγκέντρωση της ποσοστώσης, την αιρεσιμότητα. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για αυτά τα τέσσερα θέματα μέσα στο πλαίσιο των κανονιστικών μέσων. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Ρίκα Μάνερ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά τα τέσσερα σημεία, γιατί μιλήσαμε για τα θέματα αυτά με τον ε, Επίτροπο προηγουμένως, κυρίως για το θέμα της ευελιξίας για τις ποσοστώσεις. Όσον αφορά για την εδαφική συνεργασία, όπως είπε και ο Επίτροπος, χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Για τα θεματικά θα έλεγα σίγουρα, αν σταθούμε εμεί σε τέσσερις μόνο θεματολογικές ε, προτεραιότητες ε, δεν θα αντιμετωπίσουμε με τίποτα τις ε, προκλήσεις ε, των διασυνοριακών περιοχών και στις μεταφορές αλλά και τη δημογραφική πρόκληση ή θα προσθέσουμε θεματολογικές προτεραιότητες 4 ή 5 ή αλλιώς θα διευρύνουμε την ευελιξία. Υποστηρίζω πάντως ό,τι έχει γράψει ο εισηγητής σχετικά για το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή. Δεν θα πρέπει να δώσουμε ειδικά κονδύλια για το ΦΕΣΡΑ 52% όπως υπόθηκε. Εγώ συμφωνώ με την Κωνστάνς όταν, λέει, όταν μιλάει για την απασχόληση Πώς είναι δυνατόν εμείς να δημιουργήσουμε κίνητρα για την απασχόληση διότι το μέσο μπορεί κάλλιστα να αλλάξει μέρα με τη μέρα. Σε μια περίπτωση μπορεί να είναι ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή μετά να γίνει κάτι άλλο. Το κοινοτικό μέσο στη χώρα μου λειτουργεί προσθετικά με τα εθνικά μέσα θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα σε όλους τους τομείς με τα κράτη-μέλη. Για τις κατηγορίες σημείο 5 και τις περιφέρειες. Εγώ έχω διαφορετική θέση από τον εισηγητή. Δεν συμφωνώ με την ε, μεταβητική ή μη μεταβατική περίοδο και το εξήγησα ήδη. Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένα νούμερα. Τι σημαίνουν όλα αυτά και πόσο θα στοιχήσουν στο τέλος. Και μετά η μεταβατική περίοδος δεν είναι καθόλου μα καθόλου διαφανής. Τώρα για την απλούστευση εμείς συζητήσαμε αρκετά σήμερα για την περιφερειακή συνεργασία. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συμφωνώ με το καταποκοπήν 50% ε, και ένα άλλο στοιχείο της απλούστευσης θα ήταν η αναρμόνιση της συγχρηματοδότησης για όλες τις χώρες. Υποστηρίζω θερμά αυτό το σημείο γιατί ξέρω ότι στο μέλλον θα γίνει μεγάλη συζήτηση. Είναι όμως πολύ σημαντικό να έχουμε μία σαφή γραμμή. Η απλούστευση πρέπει να γίνει και σε επίπεδο βάσης στη βάση δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν όλα αυτά τα, τα, χαρτιά. Είδα εκπροσώπους, το συνάντησα εκπροσώπους των περιφερειών και υπήρχε μεγάλη επιφύλαξη ε, εκ μέρους των ενδιαφερομένων που συμπληρώνουν αυτά τα ερωτηματολόγια. Ε, διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Θα έπρεπε, υπάρχουν διαφορές για τις επιπτώσεις. Ε, εγώ δεν... Ε, δεν είμαι τόσο επικριτική με το έγγραφο όσο οι όπως είπε και ο Λάμπερτ, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα νούμερα από την Κομισιόν και μόνο τότε θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Αλλά δεν θα το απέριπτα αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν κατά βάθο ε, θετικά χαρακτηριστικά για την αιρεσιμότητα. Εγώ συμφωνώ σε αυτά τα οποία προτείνουν εξάντια για αιρεσιμότητα εξάντε. Θα... θα ήθελα να μιλήσουμε για τις τροποποίησεις στον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές ομάδες δια ε, ε, περιφερειακής συνεργασίας. Αυτοί που ήδη έχουν φτιάξει ένα τζέκτ το χρησιμοποιούν ήδη στην καθημερινότητά τους ή αυτοί που το έχουν σχεδιάσει είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την τωρινή πρόταση του κανονισμού. Όλα λοιπόν, όλες οι επιθυμίες των μελών των τζέκτ ή αυτών που θέλουν να λειτουργήσουν ως τέτοιοι <coughs> καλύπτονται στην πρόταση της Κομισιόν. Οι δυσκολίες βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Το πρόβλημα βρίσκεται στις αρχές οι οποίες ε, θεωρούν ε, ότι ε, γίνεται ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη επί Θα έπρεπε να αποφύγουμε λοιπόν τις εθνικές, από τις εθνικές αρχές να εμποδίσουν τη σύσταση αυτών των διασυνοριακών επιτροπών συνεργασίας. Θα πρέπει αυτές οι μονάδες, αυτοί οι οργανισμοί να μην αντιμετωπίζονται αυτόνομα αλλά να αποτελούν ένα μέσο που θα επιτρέπουν να εξυπηρετήσουμε την πολιτική συνοχής και που θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε αυτό το μέσο, διότι είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική γυτνίασης και σε άλλους ε, τομείς. Για παράδειγμα, συνεργασία με τις χώρες τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται εδώ για εξωτερικές πολιτικές, απλώς πρόκειται για συνεργασίες εκτός συνόρων. Εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε. 20 τέτοιες ε, επιτροπές περιφερειακής συνεργασίας έχουν συσταθεί μετά τον κανονισμό θα έπρεπε να τις αξιοποιήσουμε πλήρως. Η Μαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να μπούμε... Για να μπω στην ουσία και για να μην μακρηγορήσω, ήδη ρώτησα τον Επίτροπο για τη θέση του σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα όμως να επιμείνω με θέματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς και δεν ε, θα δεν, έχω παρά ελάχιστες προκαταλήψεις. Ε, ήθελα να ξέρω για το ελάχιστο ποσοστό των ε, περιφερειών. να μου πούνε οι συνάδελφοι τι σκέφτονται γι' αυτό. Θα πρέπει να βρούμε μία συγκεκριμένη, μία σαφή θέση διότι υπάρχει μία έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου συμπεριλαμβάνονται οι ποσοστώσεις. Θα έπρεπε να το συζητήσουμε το θέμα και να ορίσουμε τη θέση αυτής της Επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα της θεματικής συγκέντρωσης διότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι, όσο, όσο περιορίζουμε τους στόχους, τόσο περισσότερο χάνουμε σε αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να προλάβουμε αυτές τις ε, δυνατών ανομαλίες, ας αποφύγουμε το νέο καλούπι. Για το άρθρο 5 του Κοινωνικού Ταμείου, για τη συμμετοχή των ταμείων. Ε, ακούγοντας τη συνάδελφο από τη Γαλλικία, όταν μιλάει για την παρουσίαση και παρακολούθηση, ε, θα ήθελα εγώ εδώ να επιμείνω ε, στη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης των αυτονομιών και των αυτονομιών πέρα από, την κρατική, ε, από τον κρατικό έλεγχο που πρέπει να γίνει. Αυτά είχα να πω. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη των άλλων συναδέλφων. Τώρα θα έχουμε σχόλιο από τον Νίκολα Μάρτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι από την πλευρά της Επιτροπής ε, επικροτούμε την εργασία την οποία γίνεται. Τα έγγραφα προχωρούν. Υπάρχει μια εμβάθυνση στις θέσεις που έχουν εκφραστεί και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μια καλή βάση για το, τις μελλοντικές πιο εστιασμένες συζητήσεις για τις εισηγήσει για την κάθε μια μεμονωμένα. Θα ήθελα να αρχίσω με τα τέσσερα θέματα. Πρώτα απ' όλα την θεματική συγκέντρωση και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε υπάρχει μια κοινή άποψη, κοινή γνώμη για αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Υπάρχει ανάγκη συγκέντρωση, αλλά και ανάγκη ευελιξία. Δεν θέλουμε συγκέντρωση που να οδηγήσει σε ε, δυσμενή αποτελέσματα που ε, να αναγκάζει τι ε, περιφέρειες να ξοδεύουν χρήματα χωρί κανένα νόημα. Έχουμε λοιπόν μια κοινή άποψη του τι θέλουμε να επιτύχουμε και πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο μηχανισμό για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα τα μηχανισμοί είναι διαφορετικοί για τα διάφορα ταμεία. Για το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη. έχουμε έναν μηχανισμό που συνδέεται με ποσοστά. Ίσως σας φαίνεται ότι αυτή η μέθοδος είναι κάπως απλοϊκή και προσπαθήσαμε να βρούμε διάφορου τρόπους. Αυτό που μπορούμε να δούμε θεωρητικά είναι ο ιδανικός τρόπος, ε, δηλαδή να αποφύγουμε ε, να έχουμε μία λύση για όλα και να έχουμε ε, λύσεις προσαρμοσμένες, διότι αν έχουμε πλήρη ευελιξία και αν τα πράγματα για κάθε περίπτωση δεν θα έχουμε μια συνεκτική απάντηση που και αυτό βασίζεται από προηγούμενες ασκήσεις. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κάποιους περιορισμούς όταν έχουμε αυτή την άσκηση διαπραγμάτευσης. Πρέπει να έχουμε ε, σταθερές παραμέτρους ε, στην διαπραγμάτευση που ίσως επιβάλλουν κάποιο άχθος, διότι αναγκάζουν να γίνουν ορισμένες δύσκολες επιλογές, αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Θα ενδιαφερόμαστε για ορισμένες επιλογές και να τις εξετάσουμε, να δούμε αν μπορούμε ε, να προσαρμόσουμε κάτι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ορισμένοι περιορισμοί στην, στον κανονισμό θα απαιτηθούν για τους διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο από την άποψη της ευελεξίας να θυμηθούμε ότι για τα ποσοστά του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ε, σε επίπεδο εθνικό και όχι σε επίπεδο περιφερειακό. Υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ανάμεσα στις περιφέρειες ενός κράτους μέλους λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προτεραιότητες και ανάγκες. Και αυτό ισχύει διότι και οι ποσοστώσεις αναφέρονται στα ελάχιστα του κοινωνικού ταμείου και για την κατηγορία των περιφερειών σε κάθε κράτος. Αυτό επιτρέπει ευελιξία. Αλλά και ο ίδιος ε, συλλογισμός ε, ισχύει και για τα ελάχιστα ποσοστά και μερίδια του κοινωνικού ταμείου σε σχέση με την ανάγκη επενδύσεων από το κοινωνικό ταμείο στο ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και απασχόλησης και αυτό το βλέπουμε ότι είναι αναγκαίο εφόσον έχουμε αυτό το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία για τις ανάγκες. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα σε σχέση με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τις μεγαλύτερες δυνατότητες επένδυσης και περισσότερη ένταξη και ολοκλήρωση. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό το ρυθμιστικό πακέτο είναι περισσότερη ολοκλήρωση, κάτι που χάσαμε στην τρέχουσα περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί αυτή η άποψη. Και αυτό σχετίζεται με τα ε, ελάχιστες μερίδες για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μετά, για το θέμα της απλούστευσης. Χαιρετίζω το feedback από την κυρία Κρέλ για αυτό που έχουμε στον κανονισμό. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί με αυτό που συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, διότι εκεί βρίσκονται οι βασικές πρακτικές συνέπειες για τους δικαιούχους. Και ένα από τα στοιχεία που θέλω να τονίσω είναι η συνοχή, η ηλεκτρονική συνοχή, διότι είναι από τα μεγάλα ωφέλη αν τα κράτη-μέλη θέλουν να θεσπίσουν τα συστήματα που θα επιτρέπουν όλες τις επικοινωνίες ανάμεσα στους δικαιούχους και στις αρχές να γίνονται με τρόπο ηλεκτρονικό. Θα πρέπει να είναι μια υποχρέωση που θα υλοποιηθεί. Και Επίσης είναι χρήσιμο για να αποφευχθεί αυτό που λέμε gold plating σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης τα κράτη να συγκεκριμένα να υποδείξουν πώς θα μειώσουν το, το διοικητικό βάρος για τους δικαιούχους και με μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα πρέπει να περάσουν σε λεπτομερείς δράσεις και μέτρα ε, σε εθνικό ε, επίπεδο. Σχετικά με, το, με την ετήσια έκθεση πρόοδου, ε, η κυρία Κράους έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που θέλουμε είναι μια, ένα βασικό σύστημα αναφορών που συμπληρώνεται με μια λεπτομερή ανάλυση και αυτό είναι το βασικό σημείο. Ε, νομίζω ότι η κανονική αναφορά η αιτήσια θα πρέπει να είναι μια τακτική διαδικασία που προέρχεται από την παρακολούθηση, από την εποπτεία και νομίζω ότι δεν είναι ένα μεγάλο βάρος, είναι μια διαβίβαση στοιχείων ε, και πάρα πολλά μπορούν να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά με τυποποιημένο τρόπο και ε, και σε δύο σημεία έχουμε την πραγματική λεπτομερή ανάλυση όπου οι υπεύθυνε αρχές μας δίνουν συμπεράσματα για το πώς πιστεύουν ότι προοδεύει ε, το πρόγραμμα. Έτσι θα έχουμε μια καλή ισορροπία ως προς τις πληροφορίες που θα έχουμε. Σχετικά με τις αρεσιμότητες, κάτι ε, για την μακροδημοσιονομική αρεσιμότητα για την οποία υπήρξε ήδη ανταλλαγή απόψεων είναι σημαντικό να δούμε τις λεπτομέρειες της πρότασης Κομισιόν. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο έχει τώρα μια πύχηση σε σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ένα μηχανισμός πυροδότησης για την ανασκόπηση των προγραμμάτων και συμβάσεων εταιρική σχέση όταν τα απαιτούν οι περιστάσεις. Και βλέπουμε ότι τώρα ότι έχουμε μια κρίση, ειδικέ ανάγκες, υψηλή ανεργία των νέων, αυτός ε, είναι ο εκπυρσοκροτητής που θα μας επιτρέψει να κάνουμε μια ανασκόπηση και να δούμε αν χρειάζεται αλλαγή διότι οι ε, συνθήκες έχουν αλλάξει από την αρχή του προγράμματος και είναι το πρώτο μέρος ε, αυτό που ονομάζουμε ρεσιμότητα μακροδημοσιονομική, ένας μηχανισμός πυροδότησης για το μήπως ε, νέα προσαρμογή του προγράμματος. Μετά το δεύτερο ε, στοιχείο μπορεί να προκαλέσει αναστολή. Ε, είναι, αυτό σχετίζεται με την κατάσταση όπου ένα κράτος έχει αποτύχει να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις για δράσεις που θα πρέπει να καλύψουν ελλείμματα και ανισορροπίες. Ο συλλογισμός εδώ είναι απλός. Αν ένα κράτος μέλος συστηματικά έχει αποφύγει να δράσει ε, και έχει θέσει σε κίνδυνο όχι τα όσα συμβαίνουν στο ίδιο το κράτος του, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης δεν θα ε, πρέπει να αφαιθεί έτσι ως έχει. Θα πρέπει κάτι να γίνει και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται χρήματα σε αυτό το κράτος μέλος. Αλλά υπάρχει βεβαίως διακριτική ικανότητα στην κρίση του τι συμβαίνει για να δει κανείς ποια είναι η σοβαρότητα της κατάστασης, αν επαναλαμβάνει αποτυχίες και αστοχίες στο κράτος μέλος, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει αναλογικότητα. Μετά σχετικά ε, με το δεοντολογικό κώδικα που αναφέρθηκε, διότι είναι σημαντικό να πούμε ότι παράλληλα με αυτά που προετοιμάζουμε για το CSF, για τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε να είναι διαθήσιμα για να δείτε τις ιδέες της Κομισιόν, το κάνουμε το ίδιο με το δεοντολογικό κώδικα και αυτό επίσης θα μπορεί να είναι ένα άτυπο έγγραφο που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία. Ο χρονοδιάγραμμα θα είναι παρόμοιο και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο τέλος του Φεβρουαρίου ή λίγο χρόνο μετά το τέλος Φεβρουαρίου. Μετά ίσως θα πρέπει να επανέλθω ε, στο μέσο Connecting Europe, ε, πάρα πολύ σύντομα όμως νομίζω ότι αυτό που ε, πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με τα κονδύλια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε αν υπάρχει αποτυχία. Γι' αυτό υπάρχουν τρύπε, ε, γι' αυτό υπάρχουν, ε, δεν έχουμε τις πλήρεις διαμεθοριακές συνδέσεις για τα δέκα διευρωπαϊκά δίκτυα όταν έχουμε χρήματα για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, το κράτος μέλος αποφασίζει πώς θα ξοδευτούν τα χρήματα αυτά και ίσως το κράτος μέλος δεν θέλει να κάνει τη διασύνδεση διότι δεν βλέπει άμεσο όφελος για τις προτεραιότητες τους. Γι' αυτό ίσως υπήρξαν ε, διάφορες αστοχίες και αποτυχίες. Αν εξετάσουμε από την άποψη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τα εξετάσουμε όλα μαζί και να εστιαστούμε σε αυτήν την ιδέα pipeline αγωγού ε, για να δούμε ότι υπάρχει ε, σε ένα κράτος ε, μέλος βασικές υποδομές μπορούν να χρηματοδοτηθούν με διαφορετικούς τρόπους και τα κράτη-μέλη θα μπορούν να θέσουν προτεραιότητες ούτως ώστε ακόμα και αν υπάρχει αυτή η ιδέα, η αρχή του όποιος έρχεται πρώτος εξυπηρετείται πρώτος θα πρέπει να μπορεί όμως και το κράτος μέλος να ετοιμάσει το διάβλο ούτω ώστε σε κατάλληλο χρόνο να παρουσιάσει τα έργα ε, περιμένοντας ότι ε, θα χρηματοδοτηθούν τα έργα αυτά με βάση από το μέσο Connecting Europe οι δράσεις κλειδιά, οι κυριότερες δράσεις. Αυτό που θέλουμε πιστεύω να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την έννοια των κύριων δράσεων στο CSF για να μπορέσουμε ακριβώς να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες ποιες επενδύσεις θα καλυφθούν από τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επανέλθουμε στο μέλλον όταν το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι πλέον διαθέσιμο. Τώρα, επανερχόμενος στο ETC και την θεματολογική επικέντρωση. Εν μέρη απάντησα τις παρατηρήσεις στα θέματα που αναφέρθηκαν. Το άλλο στοιχείο κλειδί όμως που πρέπει να υπογραμμίσει κανείς είναι ότι υπάρχει μια εξειδικευμένη επέκταση που καλύπτει τις μεταφορές. Βλέπουμε τις μεταφορές σαν κάτι που έχει δυνάμει, μεγάλο δυναμικό στα διαμεθοριακά προγράμματα και η διατύπωση είναι επαρκώς πώς να το πω, ρητή άμεση μεταφορά στην διατύπωση των προτεραιοτήτων επενδύσεων για το ETC, τα προγράμματα ETC. Νομίζω αυτά καλύπτουν τα κυριότερα σημεία, έτσι. Χωρίς μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Πολλά μπορώ να κάνω, αλλά εξαρτώμαι από το Επί πόσο διάστημα θα μιλήσετε για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. I think the, Ναι, νομίζω ότι κατανόησα ότι η ερώτηση αυτή συνδέεται με το μέλλον των ε, κατηγοριών, μεταβατικών κατηγοριών των περιφερειών, προσωρινών κατηγοριών. Είναι μια νέα προσέγγιση, μια καινοτομία που εισάγεται εδώ οι πρώην περιοχές σύγκλησης ε, και οι περιοχές που δεν ήταν σύγκλησης αλλά βρίσκονται μεταξύ 75% και 90% αλλά φυσικά με μια κλιμάκωση όσον αφορά την ενίσχυση, την ένταση της βοήθειας όπως επισημάνθηκε. Και γι' αυτό λοιπόν με κάποιες διακυμάνσεις επίσης όσον αφορά την θεματολογική επικέντρωση. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα λοιπόν τέτοια συμπίκνωσης ή επικέντρωσης που λαμβάνουν υπόψη εκάστοτε το φάσμα, το εύρος αυτό καταστάσεων στις οποίες βρίσκονται ή εντάσσονται, εμπίπτουν αυτές οι περιφέρειες στις κατηγορίες και τη διαφοροποίηση της, του ποσοστού χρηματοδότησης. Αφενός πιστεύουμε ότι η έννοια, η προσέγγιση των μεταβατικών ε, περιφερειών ανταποκρίνεται στις ανάγκες και έχουμε αυτή την λογική σύνδεση της πολιτικής αυτής με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπης 2020, αλλά αποτελεί και τμήμα αναπόσπαστο σε σχέση με το συνολικό πακέτο για τη συνοχή. Περνάμε στους κοιόδης εισηγητές. Ε, κύριε Μάνης, ε, Μάνης, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος αυτός ε, σε σχέση με τους εισηγητές όπως έχει διανεμηθεί έχει δημιουργήσει αυτή την πίεση. Είμαστε πολύ πειθαρχημένοι σε σχέση με το κύριο νομοθετικό πακέτο και την ε, εξέτασή του. Τώρα όμως ε, έχουν κάποιες άλλες επεξηγήσεις που έδωσαν οι εισηγητές και έχει επεκταθεί το φάσμα. Δεν θα μακρηγορήσω πρόεδρε. Θα μιλήσω όμως με αριθμούς αριθμητικά μεγέθη και θα ήθελα η Επιτροπή να με προσέξει. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ πολύ για το έγγραφο εργασία, το δεύτερο αυτό έγγραφο εργασία που είναι πάρα πολύ καλό, διότι είναι ευρύτερο και καλύπτει πράγματα τα οποία είχαν συζητηθεί. Το δεύτερο, το δεύτερο είναι αυτό το οποίο απάντησε και είπε ο κύριος Χάν, ότι οι χώρες θα μεριμνούν για το πώς θα συμμετέχουν οι περιφέρειες. Ένα βήμα πίσω. Συγγνώμη, οι εισηγητέ όμω συνέταξαν σαφώ. Σαφή εταιρική σχέση πρέπει να προβλέπετε. Γιατί, πολύ εύκολο να γίνει κατανοητό, η περιφερειακή συνεργασία θα έχει 32% περισσότερα κονδύλια. Έχουμε λοιπόν 8,8 δις. Στη συνέχεια 11,7 δις στην άλλη κατηγορία. Η διαφορά είναι κάτι λιγότερο από τρία δί. Μπορείτε να φανταστείτε μεγάλο ομοσπονδιακό κράτο, δίπλα σε μικρό. Αν δεν δραστηριοποιηθούν ε, οι περιφέρειες δεν θα υπάρχει τέτοιου είδου συνεργασία διαμεθοριακά μεταξύ περιφερειών. Αν δείτε την απορρόφηση δεν υπάρχει καλό ποσοστό τέτοια απορρόφηση σε τέτοια προγράμματα. Γι' αυτό τον λόγο είναι θεμελιώδε ε, αυτό το οποίο αναφέρθηκε από του συζητητέ. Πρέπει να υπάρξουν καθορισμοί, προσδιορισμοί τι θα δοθεί σε ποιον λαμβάνοντας υπόψη την ελαστικότητα και τις ποσοστώσεις. Αυτό είναι καινούριο. Αν δούμε την έκθεση Μπάρκης, αναφέρονται τρεις-πέντε προτεραιότητες και αυτό που είπε ο κύριος Αν, τουλάχιστον τρία πράγματα πρέπει να διασφαλίζονται. Έρευνα, διαμεθοριακή αντιμετώπιση της ανεργίας και ε, σε σχέση με αυτή, ε, ε, την προσαρμογή σε σχέση με τους στόχους της ανάπτυξης. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πούμε τόσο εύκολα ότι χρειάζονται περισσότερα, διότι μπορούν εύκολα να δοθούν παραδείγματα χωρών που έχουν δώσει πολλά κονδύλια 20-50 χρόνια πριν με διαφορετικούς τρόπους για καλές υποδομές και όλα αυτά αλλά όχι για τις επιχειρήσεις στο τέλος τέλος και βλέπουμε ότι βρίσκονται σε προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τέτοιες χώρες και υποστηρίζονται πλέον βοηθούνται επειδή αντιμετωπίζουν χρεοκοπία δεν έτσι κατονομάσω αλλά είναι γνωστό το τι συμβαίνει για αυτούς τους λόγους πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό με την Επιτροπή όσον αφορά προτεραιότητες όσον αφορά την ελαστικότητα δεν είναι εύκολο να πει κανείς ε, ε, ότι α, δεν γίνεται τίποτα άλλο, πρέπει να είμαστε πάντα ανεξάρτητοι για τη Βαλτική ε, και σε σχέση και με τη Μεσόγειο. Λοιπόν, το δεύτερο αφορά τις κατηγορίες περιφερειών. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά είναι να μην υπάρχει ζήλια, φθόνος, να μην φθονεί ο ένας τον άλλο. Διότι, προσέξτε, αριθμοί, τι λένε, αν αποκλείσουμε το μέσο διασύνδεσης για τις μεταφορές η πολιτική συνοχή θα έχει 17 δις λιγότερα τα επόμενα 7 χρόνια είναι μείον 4,1%. Αν πάρουμε αυτό το μέσο για τις μεταφορές και το προσθέσουμε θα είναι 6% παραπάνω. Θα σημειωθεί αύξηση. Αλλά κοιτάξτε πρέπει να δοθεί μάχη. Δηλαδή Παρασκευή βράδυ να ξεκινήσει μία εκ των άνω προς τα κάτω προσέγγιση και ξέρουμε ότι όπως είπε ο Λεβαντόφσκι μια τέτοια προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω σημαίνει περικοπές. Και θα πρέπει εδώ να δοθούν επεξηγήσεις για αυτές τις περικοπές. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν πρόσθετα κονδύλια, θα γίνουν περικοπές είναι καθόλου εύκολο αυτό. Και όσον αφορά τι περιφέρειε, αυτό που χρειαζόμαστε ω απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει λέει φθόνο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα γιατί συμμετέχουμε εμεί ω χώρε. Η μία χώρα ω χώρα συνοχή, η άλλη ω μεταβατική χώρα ή μεταβατικών περιφερειών, η άλλη αντι, ε, ανταγωνιστική χώρα ή ανταγωνιστικών περιφερειών. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τι θα γίνει ανακεφαλήν στην διάθεση των κονδυλίων ανακεφαλήν. Αν ο αριθμός των κατοίκων που θα βρίσκονται στη μεταβατική περίοδο, ε, κατηγορία περιφερειών και έχουμε και το phasing in, phasing out, τότε τα κονδύλια είναι ανώτερα. Όμως το 47% δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αυξηθεί, θα αυξήσει τον αριθμό των πολιτών, των κατοίκων αυτών των περιφερειών. Λοιπόν, σε σχέση με τις μεταβατικές αυτές περιφέρειες πρέπει να δοθεί σαφής, αναμφίσιμη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί και ευμενείς και να μας δώσετε τελικά κονδύλια σε σχέση με ανακεφαλή όσον αφορά τους κατοίκους, τι θα δοθεί, τότε μπορούμε να τα δούμε καθαρά. Γιατί εδώ πληρώνονται δισεκατομμύρια λιγότερα, όμως μεταβατικές ε, περιφέρειες θα έχουν συν 47% και εκείνοι που είναι σε ανταγωνιστικές περιφέρειες θα βρεθούν όπως είπε ο Χάν στην, στην ίδια κατηγορία, μείον 2 κάτι της εκατό. Εδώ δεν έχουμε τέτοια μετάθεση σε μεταφοράς, μετάφραση των ποσών ανακεφαλήν. Οι άλλοι θα φθονούν γι' αυτό. Ο ένας θα φθονεί τον άλλο. Θα λέει ο ένας δεν αντιμετωπίστηκα δίκαια, εσύ ευνοήθηκες, πρέπει να επιληθεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει καλή δουλειά. Πρέπει να υπεξηγήσει τα πράγματα με πειθό για να γίνουν αποδεκτά. Και τα τελευταία δύο πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ε, μην βασίζεται κανείς ε, στην απλή ρύθμιση. Η περίοδος 2007-2013 είναι πολύ πιο περίπλοκη, διότι επιπλέον μέσα ελέγχου έχουν εισαχθεί για τα μεγαλύτερα σχέδια. Είναι και πιο περίπλοκη από ό,τι στο παρελθόν, το 2000 έως το 2006. Όμως ο αριθμός των σφαλμάτων, των λαθών, ε, μειώνεται σημαντικά. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις από το ελεγκτικό συνέδριο που να έχουν ανοιχνευτεί. Και είναι πλέον σαφές εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα οδηγήσει σε μια πλούστευση που να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ελαστικότητα στη χρήση των αριθμών, των ποσών. Διότι με τέτοια αύξηση θα αυξηθούν και τα σφάλματα στο τέλος τέλος. Λοιπόν, παρακαλώ, προσέξτε το. Πιστεύω ότι δεν είναι λογικό να πούμε «Ωραία, δώστε μας λεφτά στα ίσια» και δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι και εφικτό να γίνει. Χρειάζεται σε βάθος ανάπτυξη ε, εξέταση να δούμε πώς μπορούν να πλουστευτούν οι διεργασίες. Και τώρα, όροι και προϋποθέσεις εξάντε ή εξπόστο. Εδώ γίνεται πραγματικά παρακολουθούμε να συμβαίνει το χάος. Διαφορετικοί κανόνες και κανονισμοί. Έχουμε έξι πακέτα με τρεις κανονισμούς οικονομικών θεμάτων, ισορροπη, ισορροπημένη οικονομία και τρεις, τρεις, διατά, τρεις κανονισμούς για την δημοσιονομική πειθαρχία. Εντάξει, βαίνει καλό σε αυτό, όμως είναι υποχρεωτικοί αυτοί οι κανόνε για εκείνε τι χώρε που είναι στην Ευρωζώνη. Για εκείνε τι χώρε που βρίσκονται εκτό Ευρωζώνη δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα πλαίσια ή μπορεί και να μην ενταχθούν σε αυτά. Και τελευταίο θέμα. Αυτά τα οποία αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. 26 αρχηγεία κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν, είπαν. Συμφωνούμε μέχρι τον Ιούνιο 2012 να υπάρξουν νομοθετήματα για τη δημοσιονομική πειθαρχία και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και το θέμα της, ε, των δημοσιονομικών ελλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Προσέξτε, το ζήτημα είναι αν δεν είναι αυτά υποχρεωτικά τα πακέτα αυτά σε σχέση με τις κυβερνήσεις. Ακόμα και μετά τις προσαρμογές των νομο, της, της νομοθεσίας υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα κράτη της ζώνης ευρώ, αυτό θέτει πολύ μεγάλα ζητήματα. Αν προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέσει όρους και προϋποθέσεις για εταιρικές σχέσεις ε, εξ πώς τη όρους και προϋποθέσεις μόνο για την πολιτική συνοχή, τότε αν κάποιος είναι εκτός Ευρωζώνης, όλοι αυτοί οι νόμοι δεν είναι υποχρεωτικοί, δεν είμαι υποχρεωμένος να ε, συμμορφώνομαι. Θέλω όμως να αποτελώ μέρος της πολιτικής συνοχής και τότε θα πρέπει να μπορέσω να συμμετέχω. Πρέπει όμως αυτά να είναι αναμφίσιμα. Δεν μπορεί κανείς να μπαίνει από την πόρτα ή από το παράθυρο. Το θέμα είναι ότι εδώ υφίσταται πρόβλημα για το διαφορετικό καθεστώς των διαφορετικών χωρών. Είτε θα είμαστε όλες χώρες πολιτικής συνοχής ή όχι. Δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε διαφορετικά πλαίσια για εκείνους που είναι στην Ευρωζώνη, εκείνους που είναι εκτός Ευρωζώνης. Είμαστε όλοι μέλη όσοι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία της πολιτικής συνοχής. Δεν μπορούμε να κατακαιρματιζόμαστε διαφορετικά. Δεν γίνεται παρά αυτή η απόφαση που ελήφθη το Δεκέμβριο από του αρχηγού κατών και κυβερνήσεων μέχρι τα μέσα αυτού του έτους πρέπει να μεταφραστεί με συνεκτικό ε, ε, με τρόπο που θα οδηγεί σε σύγκληση. Διαφορετικά θα υπάρξει χάος. Δεν θα κατανοεί κανείς τι είναι υποχρεωτικό και τι όχι και με τι θα συμμορφώνεται. Και αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι δεν βρήκα τη βάση επί του οποίου θα μπορούσε ο κύριος Ρεν να πει ότι ίσως θα αφαιρεθεί από την Ουγγαρία ένα τρει. Πήραν 1,2 δις, 85% θα αφαιρεθεί. Δεν βρήκα τη νομική βάση για να γίνει κάτι τέτοιο. Και είπε ο κύριος ε, Χαν, δεν θα γίνει αυτό το 2000, ε, παρά το 2014. Αν το 2013 ε, αναφέρεται για τις πληρωμές, δεν βρήκα καμία βάση γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διαφορετικά θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Η νομική βάση είναι ο γενικό κανονισμό που υφίσταται, λέει η πρόεδρο, για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχή. 85% να αφαιρεθούν κονδύλια από μια χώρα. Όχι, αυτό δίνει μια δυνατότητα. Δεν ακούγεται η παρέμβαση του ομιλητή του μέλους χωρίς μικρόφωνο. Έχουμε τώρα λίγο χρόνο να ε, παρέμβουν οι υπεύθυνοι για να απαντήσουν στι ε, τοποθετήσει του κυρίου Μάρτιν. Κορνέλια Ένστ παρακαλώ έχει τον λόγο. Ναι, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε σε τρία λεπτά. Η ομάδα μας δεν είχε ευκαιρία παρά μόνο ελάχιστα να παρέμβει. Λοιπόν, θα ήθελα για αυτό το έγγραφο να πω για τους δύο εισηγητές, η Κωνσταντσε Κρέβ και για τον Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι, αυτά τα οποία παρουσίασαν επ' αυτόν πρώτον, μέσω των delegated acts πρέπει πολύ νυφάλια και ήρεμα να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι πού θα εφαρμόζονται και πού όχι αυτές οι προτάσεις στο συνολικό πακέτο των κανονισμών. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται να ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Το θέμα το οποίο τέθηκε εδώ σε σχέση με το έγγραφο εργασία, θέλω να το απαντήσω. Είμαστε υπέρ τη πρώτη εναλλακτική λύση που προτάθηκε, δηλαδή σε σχέση με την νομοθετική διεργασία. Δεύτερη σκέψη, εταιρικέ συμφωνίε. Το θέμα των εταιρικών συμφωνιών πρέπει ξεχωριστά να το εξετάσουμε. Δεν είναι σαφέ ποιο θα είναι εταίρο, κατά πόσον θα είναι δεσμευτικέ αυτέ οι συμφωνίε, ποιο χρονικό διάστημα θα προβλέπετε για αυτέ. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, πιστεύω, με τα λειτουργικά προγράμματα να τα περάσουμε όλα συλλήβδην και ισοπεδωτικά σε ένα πλαίσιο Τώρα, για τη θεματολογική επικέντρωση, να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Για ποιο λόγο θέλουμε να υπάρχει αυτό. Έχουμε θεματολογικούς στόχους που περιγράφονται. Γιατί χρειαζόμαστε τώρα προτεραιότητες Στοχοθετημένε προτεραιότητε, τι χρειαζόμαστε για να αποφευθεί η κατάχρηση. Τις χρειαζόμαστε διότι θέλουμε κάποια κεντρικά σημεία πολιτικά θέλουμε να προαχθούν. Γιατί χρειαζόμαστε θεματολογική προσέγγιση. Αν αποσαφηνίσουμε όλου αυτού του όρου που προανέφερα δεν, χρειάζον, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό είναι εκείνο που πρέπει να ρυθμιστεί Ποσοστώσει. Το βλέπω και εγώ όπω και οι δύο εισηγητέ αυτό το θέμα των ποσοστώσεων. Ο αυστηρό επιμερισμό ή προσδιορισμό ποσοστώσεων δημιουργεί προβλήματα και όσον αφορά και το συσχετισμό του ESF Τώρα, για το 25% το οποίο ανέφερε η Κωνσταντσε Κρέλ ως ελάχιστο, το οποίο μπορεί κανείς να το ξεπεράσει, μπορώ να το δεχτώ. Όλα τα άλλα όμως δημιουργούν προβλήματα. Όροι και προϋποθέσεις. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Γιατί να πληρώνει μια περιφέρεια την κατάσταση ότι δημιούργησε προβλήματα ένα κράτος μέλος σε αυτή την περιφέρεια με τη στάση του. Αυτό δεν, εποφε... δεν ωφελεί ούτε την περιφέρεια ούτε κανένα. Δεν φταίει η περιφέρεια για αυτά τα οποία πήγαν στραβά από την κρατική, την κεντρική κυβέρνηση του κράτους και πρέπει να δούμε και σε σχέση με τους όρους και οι προϋποθέσεις εξ άντε που είναι μαζική όρη και προϋποθέσεις είναι πραγματική απειλή. Απειλή είναι για εκείνους που θα είναι αποδέκτες των κονδυλίων και θα πρέπει να υποφεληθούν από αυτά. Ε, πρέπει να προβληματιστούμε λοιπόν για όλα αυτά, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Άλλο ένα θέμα, μεταβατικές περιφέρειες. Μεταβατικές περιφέρειες μάλιστα χρειαζόμαστε αυτή την ενδιάμεση μεταβατική κατηγορία, αλλά να δούμε πάλι τι γίνεται με αυτές. Να μην είναι μια θεά μάζα, μια γκρίζα ζώνη, έχουμε και διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών αυτής της μεταβατικής κατηγορίας. Και πολύ σωστά αναφέρεται και πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι διαφορές, ποιες περιφέρειες είναι αυτές, από πού προέρχονται και πώς χαρακτηρίζονται, ποιες είναι οι, τα στατιστικά, ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία και οι επιπτώσεις που δημιουργούνται και οι συνθήκες στις κατηγορίες, ε, για παράδειγμα πάνω από 75% νομίζω πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε απλούστευση, δηλαδή διαπίστευση, διαπίστευση όσον αφορά ε, είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται θα έλεγα και για τους ετήσιους λογαριασμούς. Ετήσιοι λογαριασμοί, και αυτοί μπορούν να συνδεθούν με υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος ως επιβάρυνση. Τελευταίο σημείο, ελαστικοποίηση, ευελιξία. Όταν κάνουμε λόγο για τη χρηματοδότηση πρέπει να επεκταθεί η έννοια της ελαστικότητας και όχι να συρρυκνωθεί, να μειωθεί. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να τοποθετηθεί σε αυτές. Ευχαριστώ τώρα. Ο, ο Μιχαήλ Τρεμόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συνάντηση με τους οικειώδεις εισηγητές. Ε, εμείς ως πράσινοι συμφωνούμε ε, με τον εισηγητή. Είμαστε άλλωστε εναντίον των μακροοικονομικών όρων. Θα ήθελα να αναφέρω και άλλα στοιχεία, όπως το αποθεματικό επίδοσης που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε μια καλύτερη ποιότητα των προγραμμάτων. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ. Σχετικά με τη διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης αν και οι περιφέρειες θα έχουν 10 ε, δισεκατομμύρια λιγότερα στη διάθεσή τους, αυτό είναι αποδεκτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζει τα προγράμματα πιο αποτελεσματικά και έτσι θα τρέξουν καλύτερα. Όσον αφορά το νέο σημείο, σχετικά με την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων πάνω στη θεσμική ικανότητα είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμφωνώ με πολλούς από τους προλαλήσαντες συναδέλφους και δεν θα ήθελα να επαναλάβω τίποτα. Τώρα Αναρωτιέμαι με την εμπειρία του παρελθόντος ότι δεν χρειάζεται να έχουμε αυστηρές ποσοστώσεις ή θεματικές ε, ε, ενότητες. Θα έπρεπε να ορίσουμε ένα ελάχιστο ποσοστό και οι χώρες να μπορέσουν να διασφαλίσουν μία αυτονομία για να ορίσουν τους στόχους τους και αυτό και για να καλύψουμε και τα ζητούμενα μέσα από τη στρατηγική 2020. Για τα γενικά σχόλια τώρα θα πω ότι συμφωνώ με προλαλήσαντες συναδέλφους και που μου μίλησαν για τους θεματικούς στόχους. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε 11 στόχους εδώ, αυτούς τους στόχους, αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι χρειάζεται μία ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού και φυσικά θα καταθέσουμε τροπολογίες και θα τα ξανασυζητήσουμε για την προετοιμασία των συμφωνιών συνεργασία. θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και τις θέσεις της τοπικής αυτοδίκησης. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε οτιδήποτε αν δεν τους έχουμε διαβουλευτεί. Τώρα για την αναιρεσιμότητα εξάντε, αυτή η έννοια δεν έχει οριστεί σαφώς. Παρόλα αυτά, όλα αυτά μπορούν να έχουν επιπτώσεις, θα μπορούσε κάλλιστα η Κομισιόν να αποφασίσει να αποφασίσει να άρει τις πληρωμές. Θα έπρεπε κατά συνέπεια να έχουμε τις πηγές αυτών των πόρων. κυρίως όσον αφορά στα μακροοικονομικά μέτρα αλλά αυτό εξαρτάται σαφέστατα από την οικονομική κρίση η οποία αλλάζει συνέχεια τα πράγματα. και κυρίως αλλάζει τα πράγματα και δεν θα πρέπει οι χώρες, οι περιφέρειες μάλλον, να τιμωρούνται και να τιμωρούνται μέσω του κοινωνικού ταμείου. Κύριε Σταυρακάκης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, τον Λαμπέρτ και την Κωνσταντζα για το έγγραφο εργασίας εξαιρετική δουλειά, σαφές και ξεκάθαρες θέσεις, αλλά και εντοπισμός των σημείων που χρήζουν περαιτέρω ανάλυση και ενημέρωση. Συμφωνώ και υποστηρίζω τις θέσεις που εκφράζονται. Από τα τέσσερα σημεία που έχουν προταθεί για συζήτηση θα ήθελα να σταθώ και εγώ ιδιαίτερα στο σημείο της απλοποίησης. Η απλοποίηση των κανονισμών αποτέλεσε μία από τις κύριες διεκδικήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η πρώτη δική μου ανάλυση του Γενικού Κανονισμού βεβαιώνει την αρχή ότι η απλοποίηση είναι πολύπλοκη διαδικασία. Όπως πολύ σωστά μας είπε η Κωνσταντζα στην εισαγωγή της, δεν είναι ξεκάθαρο αν οι προτάσεις για απλοποίηση ανταποκρίνονται στις δικές μας προσδοκίες, αλλά και στις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτικής συνοχής. Πέρα όμως από τα θέματα που αναφέρονται στο έγγραφο, εργασίες και με τα οποία συμφωνώ απόλυτα, θα ήθελα να θέσω δύο ακόμα θέματα. Πρώτον, μία από τις προτάσεις για απλοποίηση το 2008 ή 2009, αν θυμάμαι καλά, ήταν αντί η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συμφωνούν στο 100% των προγραμμάτων, η συμφωνία να γίνει στα κύρια σημεία του partnership contract, ώστε αυτό να είναι πλέον εντό εισαγωγικών ελαφρύ, μειώνοντα σημαντικά την γραφειοκρατία και τα κράτη-μέλη να διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξία στα υπόλοιπα μέρη του. Θα παρακαλούσα την Επιτροπή να μας ενημερώσει αν εξέτασε αυτή την πιθανότητα. Και τέλος, το δεύτερο σημείο είναι η πρόταση του κανονισμού επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση των τριών ταμείων της πολιτικής συνοχής σε επίπεδο επιχειρησιακών πραγμάτων, αλλά όχι σε επίπεδο αξώνων προτεραιότητας, priority axis, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις του κοινωνικού ταμείου. Θα παρακαλούσα επίσης την Επιτροπή να μας ενημερώσει αν εξέτασε την πιθανότητα αυτή. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκολας Μάρτιν τώρα δεν έχετε βεβαίως πάρα πολύ χρόνο διότι έχουμε και τους δύο εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος σχετικά με τα βασικά θέματα που τέθηκαν. Νομίζω ότι θα αρχίσω με μερικά σημεία για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Εδώ είναι σημαντικό ε, να θυμηθούμε ότι ε, οι τομείς του προγράμματος ε, πρέπει να υιοθετηθούν από απόφαση της Επιτροπής. Είναι μια διαδικασία που που συνεχίζεται, δεν μπορεί να γίνει από τα κράτη. Τα, προγραμματική τομής για τα προγράμματα αυτά είναι ε, αυτό που θα έχουμε για το 2007-2013, αυτό που είχαμε. Αλλά θα δούμε αν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ορισμένες ρήτρε ασφαλείας. Σχετικά με τα στοιχεία ε, που ζητήσατε, θα δω αν μπορούμε να δώσουμε κάτι σαφές. Ε, δεν έχω κάτι σήμερα ίσως διμερός αν θέλετε θα, ε, να, μπορούμε να δούμε αν σας δώσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε όλους. Θα, βεβαίως θα είναι στοιχεία που θα δώσω στην Επιτροπή. Για την απλούστευση δεν θα πρέπει κανείς να την παρουσιάσει ως αντίφαση Αντίθετα, θα πρέπει να δούμε την απλούστευση ως έναν μηχανισμό για την επίτευξη μείωση των σφαλμάτων, κυρίως ως προς τους κανόνες επιλεξιμότητας. Αν έχετε σαφείς κανόνες που είναι εναρμονισμένοι, θα είναι ένας τρόπος μείωση των κινδύνων, να, του κινδύνου να υπάρξουν σφάλματα, διότι υπάρχουν λάθη και σφάλματα που γίνονται επειδή δεν υπάρχει καλή κατανόηση. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους στόχους, να μειώσουμε τα λάθη. Περνώντας τώρα στην ε, θεματική συγκέντρωση. Γιατί θεματική συγκέντρωση. Απλώς ε, επειδή η πείρα μας δείχνει ότι αν προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα δεν επιτυχάνουμε τίποτα. Πρέπει να εστιάσουμε την χρηματοδότηση και το επίπεδο εστίασης θα πρέπει να αντανακλά τον όγκο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αντίκτυπο, επιπτώσεις, αποτελέσματα αυτός είναι ο συλλογισμός και ο ε, συλλογισμός ε, για τις αιρεσιμότητες ε, εξάντε είναι να δούμε αν έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αν δεν τις έχουμε αυτό επηρεάζει αρνητικά τις ε, επενδύσεις που πηγαίνουν προς τα κατάντη. σχετικά με το cross-financing, ο λόγος για τον οποίο έχουμε μειώσει το ποσό ε, δηλαδή είναι να χρησιμοποιούνται ε, ε, από το EDF χρήματα που κανονικά προέρχονται από το κοινωνικό ταμείο. Εφόσον μπορούμε να έχουμε προγράμματα από πολλαπλά ταμεία, είναι καλύτερα να εντάξουμε τα δύο σε ένα άλλο ταμείο ένα, μια ε, μοναδική δράση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διαφορετικά ταμεία και ε, από διαφορετικά προγράμματα. Έχουμε άλλες ε, πηγές για να επιτύχουμε την ευελιξία που κρίνουμε ωφέλιμη. Σχετικά με την εξάντε αιρεσιμότητα, και εδώ και πάλι έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες στον κανονισμό στο παράρτημα 4 συμπεριζόμαστε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα που να είναι λειτουργικό. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο ούτως ώστε η πολιτική ε, να εστιάζεται περισσότερο στο αποτέλεσμα, στην επίδοση. Θα πρέπει όμως να έχουμε και καλή ισορροπία, να έχουμε ε, ευκρινή κριτήρια τα οποία να αξιολογούνται αντικειμενικά στα κρατημέλη και μετά από την ίδια την Επιτροπή. Νομίζω ότι στις επόμενες συζητήσεις με τη Δανική Προεδρία και εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι νομίζω ότι μπορούμε να δούμε με ποιους τρόπους θα κρατήσουμε τα ουσιαστικά σημεία αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Όσο προς τις διαδικασίες για τις συμβάσεις εταιρική σχέσης και τα προγράμματα, εδώ και πάλι θέλουμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στο να έχουμε έγγραφα που επιτυχάνουν τους σκοπούς τους ε, που δεν είναι βαριά έγγραφα, αλλά θέλουμε κυρίως ε, να εξετάσουμε τρόπους με τα προγράμματα για το πώς μπορούν να τροποποιηθούν όταν αυτό απαιτείται και να έχουμε μια πιο ελαφριά διαδικασία από ό,τι τώρα και να δούμε τρόπους με τους οποίους το κείμενο μπορεί να προσαρμοστεί για να επιτευχθεί αυτό και θα πρέπει και να δούμε τρόπους και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για να μην υπάρξει ε, διπλή χρήση ή επικάλυψη. Σε σχέση με, την, με τις προτεραιότητες, ο βασικός σκοπός με την δομή ε, των προγραμμάτων και των αξώνων προτεραιότητας είναι να κρατήσουμε τη διασύνδεση ε, με, την, με θεματική και με την Ευρώπη 2020. Δεν θέλουμε λοιπόν υπάρχει μια διάλυση, μια διασπορά που να υπονομεύει τους βασικούς στόχους των όσων προσπαθούμε να επιτύχουμε. Είσαστε πολύ σύντομος. Κωνσταντσε, κάποια σχόλια και μετά ο Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι. Η Κωνσταντσε Κρέτ. Δεν θέλω να σχολιάσω σε ευρύ πλαίσιο. Κάποια θέματα νομίζω αναφέρθηκαν και θα παρακαλούσα. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της απλούστευσης έχει συντάξει, ε, συντάσει ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Ίσως λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Ποια είναι τα στοιχεία κλειδιά της ε, απλούστευσης ως διεργασίας και να διατεθούν αυτά ε, ως, σε ένα έγγραφο στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτό θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο για την προπαρασκευή της ακρόασης που θα έχουμε. Παρακαλώ μελλοντικά ίσως, μελλοντικά την συζήτηση να την διεξάγουμε με βάση τους επιμέρους εξειδικευμένους κανονισμούς σε μεγαλύτερο βάθος και πιο εξειδικευμένα για επιμέρους θέματα. Γιατί όταν κάνουμε κάθε φορά ένα τέτοιο μεγάλο γύρο επί παντός του επιστητού σε πολύ μεγάλο φάσμα δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Όλοι είμαστε πολιτικοί και μας ενδιαφέρουν συγκεκριμένα πράγματα. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να επικεντρωνόμαστε περισσότερο εξειδικευμένα σε κανονισμούς σε μεγαλύτερο βάθος για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, ο κύριος σας ευχαριστώ. Κάποιες σκέψεις από πλευράς μου αν θέλετε μπορώ να σας εκθέσω. Όχι μόνο να λάβουμε υπόψη από το ESF τις ιδέες αυτές που είναι γόνιμο όπως καταδείχθηκε σήμερα αλλά να έχουμε και μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της υπαίθρου να το κάνουμε αυτό με τους ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές για αυτά τα θέματα ανάπτυξης υπαίθρου διότι χρειαζόμαστε καλές ενδείξεις ε, να έχουμε θετικές ε, θετικά στοιχεία και έχω αρκετά ερωτηματικά ακόμα. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά θεματολογικά σε σχέση με τις θεματικές προτεραιότητες, τι θα γίνει με όλα αυτά. Να τα διοργανώσουμε με ένα ανοιχτό πνεύμα, πιο ανοιχτά, πιο ελαστικά και όχι μόνο μια ομάδα εργασίας. Να το κάνουμε αυτό αν γίνεται. Το ίδιο για την πολιτική για την θάλασσα, την ε, θαλάσσια πολιτική, ναυτιλιακή πολιτική για την αλληλεία. Να σας πω για την ακρόαση δύο πράγματα. Στην Επιτροπή Ήτρε έχουν ε, γουρλώσει τα μάτια τους πραγματικά. Και εξετάζουν εντυπωσιασμένοι τον στόχο 1. Γιατί αυτό. Διότι εδώ έχουμε λέει το θέμα της, ε, ε, των έκτακτων επιδόσεων, των βέλτιστων επιδόσεων και της καινοτομίας. Από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για αυτό την πρόθεση της Επιτροπής Ήτρε από κοινού να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε μια κοινή ακρόαση για αυτούς τους στόχους. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ, ας το πω έτσι, αλλά είναι και θέματα δικής μας αρμοδιότητας κάποια από αυτά. Το τελευταίο, για τη δική μας ακρόαση που θα γίνει στις 20, 20 Μαρτίου. Ίσως εδώ θα έπρεπε να συζητήσουμε με εκείνους τους ε, ανθρώπους που εμπλέκονται και έχουν πείρα διότι θα μπορούσε κανείς να έρθει σε επαφή με κάποιους μεγαλόσχημους αλλά πρέπει να πάρουμε πιο πρακτική μορφή σε αυτή την ακρόαση για να υπάρξουν άμεσα συμπεράσματα να υπάρξουν τοποθετήσεις ώστε οι συνάδελφοι να προτείνουν βελτιώσεις σε κάποιες προτάσεις και να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα μια ρεαλιστική, πραγματιστική προσέγγιση νομίζω σήμερα κάναμε κάποια πρόοδο δεν κινηθήκαμε προς κάθε κατεύθυνση επί όλου του ορίζοντα ε, Υπότιτλοι επί ε, της περιφέρειας των 360 μοιρών του ανεμολογίου. Νομίζω πρέπει εδώ να είμαστε ε, συγκεκριμένοι. Και εδώ ευχαριστούμε πολύ την Προεδρία που εισάκουσε και είπε τι είδου προγραμματισμός υπάρχει για την μία ή άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή για το ένα ή άλλο πεδίο δράσης. Το να πούμε ότι θα έχουμε μία πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο πρέπει να δούμε τι κάνουν εκείνοι από πλευρά τους. Δεν μπορούμε να διαφέρουμε εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο στο χρονοδιάγραμμά μας και τη δράση μα σε σχέση με του άλλου. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς για τον χρόνο που μας έδωσαν και παρέμειναν κοντά μας μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος με την παράταση. Υπενθυμίζω θα συνέλθουμε, θα ξανασυναντηθούμε αύριο στις 9 η ώρα το πρωί και πάλι για μια πολύ σημαντική συζήτηση και έχουμε και ψηφοφορίες αύριο, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και τον Νίκολα Μάρτιν. σας ευχαριστώ, γεια σας.